Uh, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο χρόνος περνάει, γι' αυτό παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ησυχία παρακαλώ. Καλωσορίζω εδώ τον ε, επίτροπο, τον υποδειχθέντα επίτροπο Όλη Ρεν, εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για ε, τα θέματα του υποδειχθέντος αυτού Επιτρόπου, οπότε τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα θέσουν τις ερωτήσεις αποκλειστικά σε αυτόν. Μας έχει ήδη δώσει ο κύριος Ρεν απαντήσεις γραπτά στις γραπτές μας ερωτήσεις. Έχουν μοιραστεί αυτές οι γραπτές απαντήσεις σε όλες τις γλώσσες, σε όλους τους ευρωβουλευτές. Ησυχία παρακαλώ για να ακουγόμαστε, λέει η Πρόεδρος. Ο υποδειχθείς λοιπόν ε, επίτροπος θα μιλήσει για τις αρμοδιότητές του, για την ευρωπαϊκή του δέσμευση, για την ανεξαρτησία του, για τις γνώσεις του όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει και τις ικανότητές του. Θα υπογραμμίσω λιγάκι τώρα την διαδικασία. Είναι μια γενική διαδικασία η οποία υιοθετείται από όλε τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ για όλε τι ακροάσει. Λοιπόν, μετά από τι δικέ μου παρατηρήσει, ο αποδειχτή ε, επίτροπο θα μα κάνει μια παρουσίαση δεκάλεπτη. Μετά από την εισαγωγή αυτή θα έχουμε ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές και θα ξεκινήσουμε με ερωτήσεις από έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα με τη σειρά. 32 ερωτήσεις θα μπορέσουμε να θέσουμε ως Επιτροπή από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Για την κάθε ερώτηση υπάρχει ένα λεπτό. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι μία ερώτηση κάθε φορά και δεν πρέπει να είναι ένα σύνολο ερωτήσεων, αλλιώς θα χτυπήσω το σφυρί μου. Διότι ο υποδεικτής επίτροπος θα έχει μετά δύο λεπτά στη διάθεσή του για να απαντήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι άδικο να του ζητήσετε να απαντήσει σε ένα σωρό ερωτήσεις μέσα σε δύο μόνο λεπτά. Στη συνέχεια μπορεί αυτός που έχει κάνει την ερώτηση να συνεχίσει για το ίδιο όμως θέμα, αν δεν έχει ικανοποιηθεί από την απάντηση του υποδειχθέντο επιτρόπου. Εντάξει, αν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ζητήσετε και πάλι από τον υποδειχθέντο επίτροπο να απαντήσει. Σας παρακαλώ να μην μιλάτε πολύ γρήγορα γιατί θα χάσουμε χρόνο αναγκαστώ να σας διακόψω και να σας πω να μιλάτε πιο αργά. Αν με βλέπετε εδώ με ένα κίτρινο χαρτί, αυτό να ξέρετε ότι σημαίνει ότι πάτε πάρα πολύ γρήγορα, δεν σας προλαβαίνουμε, γι' αυτό να μιλάτε λίγο πιο αργά. Δεν θέλω να διακόπτω, οπότε προσπαθήστε να το κάνετε και από μόνοι σας. Να ξέρετε ότι θα σας κόβω το λόγο όταν έχει λήξει ο χρόνος ομιλίας σας. Θα προσπαθήσω να σας προειδοποιήσω προηγουμένως, να με αυτό το κουμπάκι που κάνει πινγκ, θα πατάω το κουμπί. Άμα το ακούσετε αυτό σημαίνει ότι λίγο ο χρόνος σας και πρέπει να ολοκληρώσετε. Στο τέλος των ερωτήσεων, ο υποθέτης επίτροπος θα μπορέσει να κάνει άλλη μια δήλωση, πεντάλεπτη αυτή τη φορά. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ρεν, πάντως θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Να ξέρετε ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ εκτιμάει όλους ιδιαίτερως τις απαντήσεις σας που λέτε ότι θέλετε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα επίπεδα. Υπογραμμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα νομοθετικά και προνομοθετικά αλλά και μη νομοθετικά κείμενα, εμείς στο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, έγκαιρα παρακαλώ, προκειμένου να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε και να πάρουμε ό,τι αποφάσεις έχουμε να πάρουμε. Και μάλιστα δεν πρέπει να πρόκειται μόνο για ότι εμείς σας ζητάμε, πράγματα τα οποία εμείς ε, ρητά έχουμε πει ότι θέλουμε, αλλά και για τα πράγματα εκείνα για τα οποία εμείς μπορεί να μην έχουμε ιδέα. Αλλά εσείς να ξέρετε. Και γι' αυτά θέλουμε να φροντίσετε εσείς με δικιά σας πρωτοβουλία να μας ενημερώνετε έγκαιρα. Δεύτερον, για την μακροοικονομική πολιτική, για τα σχέδια ανάκαμψης, για τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για μας. Και τώρα στην οικονομική κρίση που βρισκόμαστε, οι αρμόδιοι επίτροποι για τα θέματα οικονομικών, νομισματικών, ανταγωνισμού κλπ. Χρειάστηκε να συνεργαστούν μεταξύ τους στενά. Η συνεργασία αυτή φανταζόμαστε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ έχει αρμοδιότητα για όλες αυτές τις πολιτικές και θέλει να συμμετέχει στην ε, ολοκλήρωση των πολιτικών αυτών και στον καθορισμό των πολιτικών αυτών. Θέλουμε όλη, ολόκληρη Επιτροπή ΕΚΟ να συμμετέχει στις διαδικασίες. Και μετά από αυτό που είπαμε πριν, πρέπει να ξέρετε ότι η Επιτροπή μας συζήτησε ήδη ότι μακροοικονομικά θέματα και οικονομικές ρυθμίσεις, δημοσιονομικές μάλλον ρυθμίσεις, δεν έχουν ε, πολύ συγκεκριμένο διαχωρισμό. Υπάρχει κάτι το οποίο συνδέει τα δύο. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια γενικά σχόλια που είχα να κάνω από την Προεδρία και ελπίζω να ακούσουμε κάτι για αυτά κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, δίνω το λόγο στον προτινόμενο επίτροπο, κύριο Όλι Ρεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Λέει στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά ο κύριος Ρεν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω τη χαρά μου για το ότι βρίσκομαι και πάλι κοντά σας, διότι κατά το χρονικό διάστημα όταν ε, ήμουν ε, Ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε ήμουν αναπληρωματικό μέλος ε, αυτής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ένας, αν θέλετε, ο σημαντικότερος κατ' εμέ ακρογωνίως λίθος της κοινωνικής οικονομίας αγοράς στην Ευρώπη. Αισθάνομαι λοιπόν ότι δεσμεύομαι από τους ε, στόχους της ε, οικονομίας αυτής. Δεσμεύομαι μάλιστα κατά ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο να αναπτυχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην οποία θα συμμετέχουν όλοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Ως εκ τούτου η συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Πρόκειται λοιπόν για τις ε, προσδοκίες των ε, πολιτών ε, στο πρόσωπό μας, απέναντι σε εμάς, κυρίως αυτή την περίοδο της κρίσης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον, θέσεις εργασίας, ευημερία, οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Κυρίες και κύριοι, ως Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος υπεύθυνο για τα οικονομικά και νομισματικά ζητήματα, επιτρέψτε μου να πω ότι ο κύριος στόχος μου είναι η ανάκαμψη, η οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς έχουμε τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε κατά προτεραιότητα, τρία εργοτάξια πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχύσουμε το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μας και ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις στρατηγικές της οικονομικής ανάπτυξης και της εξόδου από την κρίση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η νέα στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι αναγκαία προκειμένου να κινητοποιήσουμε κάθε είδους πηγές ανάπτυξης και απασχόλησης από την εκπαίδευση μέχρι τις πράσινες τεχνολογίες για να συνοδεύσουμε την Ευρώπη κατά το επόμενο στάδιο της οικονομικής της ανάπτυξης. Δεύτερον, πρέπει να σταθεροποιήσουμε τα δημοσιονομικά οικονομικά των κρατών μελών τα επόμενα χρόνια. Αυτό βέβαια απαιτεί μια αντιμετώπιση σφιχτή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των άλλων θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων στο άμεσο μέλλον. Σίγουρα η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αναγκαία όπως φαίνεται και από τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για την ανεργία, που είναι 10%, για να καταφέρουμε ε, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις, για να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία. Αλλά ε, το μέλλον των ε, δημοσίων οικονομικών, του δημοσίου χρέους, για παράδειγμα, είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας και τη δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη. Τρίτον, πρέπει να φροντίσουμε να μιλάμε με μία φωνή προς τα έξω όσον αφορά την οικονομική παγκόσμια διακυβέρνηση. Άρα πρέπει να μπορούμε να επηρεάζουμε τα πράγματα, να επηρεάζουμε τις μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών ρυθμίσεων και την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου σύντομα να σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύω να προχωρήσω για να πετύχω το στόχο μας, αυτές τις προτεραιότητες δηλαδή. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται μακροοικονομική σταθερότητα. Αλλά οι τρεις προτεραιότητες τις οποίες αναφέρομαι, δηλαδή ανάπτυξη, σταθερότητα και η ε, συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πράγματα άμεσα αλληλένδετα μεταξύ τους. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μας δίνει ένα πλαίσιο σταθερότητας των ε, δημοσιονομικών οικονομικών μέσα από μια συντονισμένη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, αλλά τα μέτρα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν όταν η οικονομική ανάπτυξη έχει επιτευχθεί. Μόνο όταν η ανάκαμψη έχει σταθεί στα πόδια της, όταν έχει ξεκινήσει για τα καλά, μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για πραγματική έξοδο από την κρίση. Έπειτα, χρειάζεται συντονισμό των πολιτικών μας. Πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός αυτός. Το είδαμε αυτό και από τα πρόσφατα γεγονότα στην Ελλάδα, τις πρόσφατες εξελίξεις. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές και του ζητάμε να ετοιμάσουν ένα πλήρες και συγκεκριμένο οικονομικό πακέτο με συγκεκριμένα και απτά μέτρα. Η κρίση έχει δείξει επίσης ότι υποφέρουμε και από ένα κενό όσον αφορά την αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου. Το προτινόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πρέπει να καλύψει το κενό αυτό. Μια άλλη προϋπόθεση για να έχουμε καλή εποπτεία είναι μια έγκυρη και άξια εμπιστοσύνης απόδοση οικονομικών στοιχείων και εθνικών λογαριασμών είναι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Ό,τι αδυναμίες υπάρχουν στο σύστημα αυτό πρέπει να διορθωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης μπορεί να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη μέσα από τη διεύρυνση της Ευρωζώνης. Κάτι για το οποίο θα δουλέψω τηρώντας βέβαια τους κανόνες και φροντίζοντας να υπάρχει ίση ε, μεταχείριση μεταξύ όλων. Μιλάμε για σταθερότητα και ανάπτυξη. Η στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 θέλει να δώσει νέο δυναμισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το, οι μηχανισμοί του συμφώνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί νέα όθηση στην στρατηγική αυτή, προκειμένου αυτή να πετύχει. Εσείς ως Ευρωβουλευτές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να πετύχει η στρατηγική αυτή. Για να συγχρονίσουμε τώρα την οικονομία μας, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να εντατικοποιηθούν οι καινοτομίες. Δεδομένων των φορολογικών περιορισμών που έχουμε, είναι δύσκολο να πετύχουμε το συνδυασμό των επενδύσεων και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ πάντως, εφόσον επιβεβαιωθεί η θέση μου στη θέση του Επιτρόπου, να ξέρετε ότι θα ξεκινήσω με την αξιολόγηση των μηχανισμών και των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και θα βάλω την Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 σαν προτεραιότητα και θα φροντίσω να υπάρξει η κατάλληλη χρηματοδότηση. Για όλα αυτά τα θέματα και για άλλες πρωτοβουλίες έχω απαντήσει στις γραπτές μου απαντήσεις. Σίγουρα είναι προτεραιότητά μου η καλή συνεργασία μαζί σας και με την Επιτροπή σας. Κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρώσω θέλω να πω, να υπενθυμίσω ότι ήμουν ευρωβουλευτής και εγώ εδώ. Οπότε και τα τελευταία πέντε χρόνια εξάλλου συνεργάστηκα μαζί σας και έχω μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σύμμαχοι και συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Η οικονομική ανάπτυξη προβάλλει Πολλέ φορές βραχυπρόθεσμα συμφέροντα. Συγγνώμη, η οικονομική ύφεση προβάλλει συχνά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα και στενά συμφέροντα. Δεν πρέπει όμως να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε να προβάλλουμε το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Με ρωτήσατε τι είναι αυτό που με κάνει να θέλω να δουλέψω σε αυτή τη θέση, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι γιατί θέλω να κάνω τη διαφορά, να δώσω νέες προοπτικές, μια ευημερούσα και δίκαιη Ευρώπη, όπως θέλετε κι εσείς. Ξέρω ότι είναι μεγάλη η ευθύνη αυτή. Το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή το οικονομικό και νομισματικό, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, ιδιαίτερα σήμερα που περνάμε δύσκολους καιρούς. Όμως θέλω να τα καταφέρω και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε εφόσον αποφασισμένα πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για μια βιώσιμη Ευρώπη. Αν δεν το κάνουμε, κινδυνεύουμε από οικονομική τελμάτωση και από πολιτικούς χειρισμούς χωρίς νόημα. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε από κοινού την ευθύνη να κάνουμε την αναγέννηση της Ευρώπης μια πραγματικότητα. Προσδοκώ καλή συνεργασία μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσει από κοινού. Ευχαριστώ. And Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο. Πρώτο ερώτημα, κύριο Γκόζη. Ζων Πολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος των μελών της ομάδας μας να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, γιατί γνωρίζετε ναι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι η πρώτη σας επίσκεψη σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και με τους συναδέλφους θα έχουμε την ευκαιρία να σας θέσουμε διάφορα ερωτήματα τα οποία θα αφορούν το γενικό πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ομά να σας ρωτήσω πώς προβλέπετε τον συνδυασμό από τη μία πλευρά της, άπετης, της απέτησης ε, υγιών δημοσίων οικονομικών που δεν είναι υποθήκη για το μέλλον και από την άλλη μεριά την πραγματοποίηση των απαραίτητων δράσεων για την έξοδο από την κρίση και την μεγέθυνση. Απάντηση. Κύριος Ρέν. Ευχαριστώ κύριε Γκοζέ για το ερώτημά σας. Είναι θεμελιώδες να υπογραμμίσουμε ότι οι δύο στόχοι, η ανάπτυξη και η έξοδο από την κρίση, δεν είναι αντίθετες μεταξύ τους. Αντίθετα, είναι συμπληρωματικές έννοιες. Μία υγιής και βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί υγιή δημόσια οικονομικά. Το υπερβολικό έλλειμμα και ένα μεγάλο χρέος υποχρεώνει τις κυβερνήσεις μας να ξοδεύουν όλο και περισσότερα μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν άλλες προτεραιότητες, παιδεία, κοινωνικές δαπάνες, έρευνα. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να επαναπροσανατολίσουμε τα δημόσια οικονομικά μας έτσι ώστε να είναι βιώσιμα για να ενθαρρύνουμε την μεγένθηση στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο για να επανέλθουμε σε υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομική ανάπτυξη και για να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο στόχους είναι απαραίτητο να αυξήσουμε την ποιότητα των δημοσίων μας δαπανών και να δημιουργήσουμε οικονομικά εργαλεία που θα συνδυάσουν την δημόσια επένδυση και την ιδιωτική επένδυση για να έχουμε τις βέλτιστες επιδόσεις και για την μεγέντηση και για τα υγιή δημόσια οικονομικά. Με αυτή τη λογική κύριε Επίτροπε τι αναμένεται από τα αποτελέσματα των εργασιών της ειδική Επιτροπής για την κρίση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή υπό την προεδρία του συναδέλφου, μου, του συναδέλφου μας κυρίου Κλίτς. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Αυτή η Επιτροπή θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο φαντάζομαι και θέλω να συνεργαστώ με αυτήν την Επιτροπή που προεδρεύεται από τον κύριο Κλίντς θα είναι σημαντικό από κοινού να βρούμε ένα μείγμα βέλτιστων πολιτικών που θα συνδυάσει βιώσιμα δημόσια οικονομικά και ταυτόχρονα επενδύσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα είναι δύσκολο έργο αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τις στρατηγικές εξόδου. Πρέπει να επαναζωογονήσουμε τα δημόσια μας οικονομικά και να βρούμε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προσβλέπω να συνεργαστώ με την Επιτροπή του, που προεδρεύεται από τον κύριο Κλίσμαν και με αυτήν εδώ την Επιτροπή θα διαδραματίσει ζωτική σημασίας ρόλο. Επόμενο ερώτημα ο κύριος Μπούλμαν, εξ ονόματος των Σοσιαλιστικού Κόμματος. Καλημέρα κύριε Ρεν και εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας. Εσείς επιδιώκετε να καταλάβετε μια πολύ σημαντική θέση σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή και θέλω να πω ότι αν δεν συμβεί κάτι το καθοριστικό, τότε στο τέλος ε, της ε, θητείας σας, την οποία επιθυμείτε να μπορέσετε να αποκτήσετε, τότε θα βρισκόμαστε ακόμα χειρότερα και πριν από το επίπεδο της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, τι είναι εκείνο που πρέπει να αλλάξουμε. Εσείς είπατε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Για δέκα ολόκληρα χρόνια εφαρμόσαμε τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πώς μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ότι θα εφαρμόσουμε εφαρμοστεί μια πολιτική που θα είναι ακόμα καλύτερη. Και πώς θέλετε να πετύχετε ότι θα έχουμε ένα νέο deal, μια νέα στρατηγική που θα, που θα είναι καλύτερη από αυτή που παρουσίασε η Κομισιόν τον Νοέμβριο, όπου απλά ήταν μια πολιτική του παρελθόντος, αυτό που απλά θα λέγαμε άλλαξε ο Μαναλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούλμαν για την ε, ερώτησή σας ε, και πράγματι θέλω να σας πω ότι και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας για το μέλλον της οικονομίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δράσουμε τώρα τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των ε, δημόσιων οικονομικών, στα δημοσιονομικά. Η στρατηγική του 2020 θεωρώ ότι θα αποτελεί ένα καθοριστική σημασίας εργαλείο σε τέτοιες εποχές, σε περίοδο κρίσης, ε, πρέπει να επιδιώκουμε ανάπτυξη αλλά και παράλληλα θέσεις εργασίας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που δίνονται να κινητοποιήσουν την οικονομική ανάπτυξη, ξεκινώντας από την εκπαίδευση, περνώντας τις καινοτομίε μέχρι και την ε, πράσινη οικονομία και τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες. Εξάλλου, πρέπει να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε το συντονισμό της ε, οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να κάνουμε καλύτερη χρήση της συνθήκης Λισαβόνας για να έχουμε καλύτερο σύστημα συντονισμού και εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δύναται να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές, να εμβαθύνουμε σε θέματα εποπτείας. Παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκδίδει συστάσεις και προδοποίησεις σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Και εγώ προτίθεμαι σύντομα να κάνω μια σχετική ανακοίνωση έτσι ώστε για να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα τόσο μεγάλη σημασία θέματα. Κοιτάξτε κύριε Ρεν, η Ισπανική Προεδρία στις αρχές του έτους πρότεινε να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση στο, στα θέματα συντονισμού και κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Εσείς τι θα λέγατε αν ανατίθετο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει τον έλεγχο της ε, θεσμικής συμφωνίας για τον πολιτικό συντονισμό και ας πούμε να προτείναμε στο Συμβούλιο ότι δεν θα υπάρχουν πλέον αλλαγές ε, στην οικονομική στρατηγική χωρίς να εισακούεται και η δική μας άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς θα συμφωνούσατε με μια τέτοια πρόταση. παρακολούθησα τη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, ε, προφανώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στη συζήτηση ε, που προκλήθηκε από την Ισπανική Προεδρία και σχολιάστηκε από διάφορα κράτη-μέλη. Κατά τη δική μου άποψη, το επόμενο βήμα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον οικονομικό συντονισμό είναι το να κάνουμε καλύτερη, μεγαλύτερη χρήση της συνθήκης της Αβώνας για να αναδιοργανώσουμε την Ευρωζώνη και θέματα εποπτείας, συντονισμό και εποπτεία. Ε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη νέα συνθήκη για να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φόρουμ. Εδώ θέλω να σας πω ότι εγώ θα εργαστώ με βάση τη συνθήκη και τη συμφωνία πλαίσιο την οποία αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμεθα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να βρούμε τους βέλτιστους δυνατούς τρόπους για να συμπεριλάβουμε το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας που θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση όχι μόνο των κατευθυντήριων γραμμών αλλά και όλων των άλλων τομέων που έχουν σχέση με την οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ερώτηση τώρα από τον κύριο Γκουλάχ. Κυρία Γκουλάχ, συγγνώμη. Και εξ ονόματος των φιλελευθέρων και δημοκρατών να σα καλωσορίσω και δίνω συνέχεια στο ίδιο θέμα. Η κρίση απέδειξε ότι όταν οργανωθήκαμε καλά, όπως κάναμε για τα νομισματικά, είχαμε ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Όταν όμως η πτυχή των οικονομικών ή της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν πιο αδύναμη, υπήρχε λιγότερη η Ευρώπη. Επανέρχομαι λοιπόν στα ίδια θέματα των ερωτημάτων που σας τέθηκαν. Τι προτείνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε η απάντηση να είναι πιο ευρωπαϊκή και όταν λέτε ότι θα εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας τι έχετε ακριβώς κατά νου. Μιλήσατε για την εκπροσώπηση προς τα έξι αλλά για θέμα συντονισμού και ακόμα παραπέρα για τον πολίτη αν αλλάξει ο όρο στρατηγική τη Λισαβόνας από το στρατηγική του 2020, γι' αυτόν τον ίδιο δεν αλλάζουν πολλά. Σας ευχαριστώ κυρία Κουλάρ για την ερώτησή σας. Τι προτίθεμαι να κάνω στον τομέα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Με δεδομένη την προχωρημένη ενσωμάτωση των οικονομιών και τα διδάγματα από την οικονομική κρίση, κατά την άποψή μου υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα για να ενισχυθεί η εποπτεία και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν και αυτά με τον στόχο αυτό. Πώς και πώς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εδώ έχω τρία να σας πω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την συνθήκη για να αναθεωρήσουμε την εποπτεία και τον συντονισμό, καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την οικονομία. Εποπτεία, παραδείγματο χάρη, η Κομισιόν θα έχει το δικαίωμα να εκδώσει συστάσεις και ε, ειδοποιήσεις. Πρέπει επίσης να κεφαλαιοποιήσουμε τα όσα έχουμε με βάση τη συνθήκη για να διορθώσουμε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και εδώ η μακροπροληπτική εποπτεία θα είναι πολύ σημαντική. Και στα πλαίσια αυτά, νομίζω ότι αυτό θέλετε ως απάντηση, στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα εργαλεία για να δώσουμε σθένος για αυτούς τους στόχους της στρατηγικής του 2020, η οποία πρέπει να παρακολουθηθεί καλύτερα και πρέπει να βασίζεται στην εταιρική σχέση και πραγματική συμμετοχή των κρατών μελών και των άλλων ενδιαφερομένων. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα από τα αδύναμα σημεία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Δεν ήταν η ιδιοκτησία των κρατών μελών. Γι' αυτό και η παρακολούθηση που έγινε μέσω του, της ανοιχτή μεθόδου συντονισμού δεν διαδραμάτισε τόσο ισχυρό ρόλο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την συνθήκη και τις κατευθυντήριες γραμμές για να δώσουμε σθένος σε αυτήν την πολιτική. Και το τρίτο μου επιχείρημα, λυπάμαι διακόπτη κυρία Πρόεδρες, έχω ένα συνεχιζόμενο ερώτημα. Ποιο είναι το τρίτο σας σημείο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ κυρία Κουλάρ. Πράγματι, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το ότι πρέπει να εργαστούμε για να έχουμε μια ενιαία εκπροσώπηση της Ευρωζώνης στα διεθνή ιδρύματα και βήματα, όπως την ομάδα των 20 ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάρο μεγαλύτερο της επιρροής μας. Γι' αυτό λοιπόν έχω την πρόθεση να σας παρουσιάσω μια ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνο για το θέμα αυτό, όταν βεβαίως το έχει συζητήσει και το Κολέγιο των Επιτρόπων. Και με αυτή τη λογική πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη, γιατί η συνθήκη δίνει τη δυνατότητα ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για τέτοιου είδους εκπροσώπηση. Σας ευχαριστούμε. Η πράσινη, κύριος Γκίγκολτ. Ja, auch von uns herzlich Herr Και εμείς ε, σας καλωσορίζουμε κύριε Ρεν. Ε, θα συνεχίσω εκεί που σταματήσατε. Δηλαδή θέλω να πω το εξή. Αν δούμε αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις, καταλήγουμε στο ότι αυτή τη στιγμή κάποια κράτη της Ευρωζώνης βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Χαρακτηρίζονται από μαζική ανεργία, από τεράστια ελλείμματα και στο άλλο τμήμα της Ευρωζώνης, αν ρίξουμε εκεί τη ματιά μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πλήρης απόκληση. Εσείς τώρα τι μας είπατε. Είπατε ότι θα εκδώσετε συστάσεις ε, και κάποιες προειδοποιήσεις. Δεν νομίζω όμως ότι αρκεί αυτό για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πιο εναρμονισμένη ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία στην πολιτική που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες που υφίστανται. Κοιτάξτε, εγώ εκτός από προειδοποίησεις και συστάσεις που αναφέρατε εσεί, δεν άκουσα να είπατε τίποτα άλλο για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ε, εγώ αναφέρθηκα ε, στη μετέρθηση της συνθήκης που κάνει λόγο για την οικονομική εποπτεία. Γι' αυτό τα είπα. Η ανεργία βεβαίως σήμερα είναι μεγαλύτερη πρόκληση και αυτό είναι τραγωδία για κάθε Ευρωπαίο που έχει χάσει τη δουλειά του με 10% ρυθμό ανεργίας, είναι αλήθεια ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να κινητοποιήσουμε όλες μας τις πολιτικές και όλες τις πηγές ανάπτυξης αυτό πάλι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους επιτρόπους, όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε κάθε ένας από αυτούς να μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Κατά την άποψή μου, αν θέλετε, η παιδεία είναι τεράστια σημασίας για να μπορέσει η, κρίση, η Ευρώπη να ε, ξεπεράσει την κρίση και να σφυριλατήσει μια πραγματική πράσινη σύγχρονη οικονομία για το μέλλον. Εξάλλου πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε καινοτομίε, χρειαζόμαστε μια λογική πράσινη ανάπτυξη. Όλα αυτά σημαίνουν ότι περιμένω πολλά περισσότερα από τους υποδειχθέντες συναδέλφους, από την κυρία Βασιλείου, από την ε, αρμόδια επίτροπο για θέματα καινοτομία, από τον κύριο Πότορσνικ, ε, που είναι αρμό θα είναι αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος. Οφείλουμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε όλους τους επιτρόπους, όλες ε, τις διευθύνσεις και τις δικές σας βεβαίως επιτροπές, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις πηγές ανάπτυξης και να καταρτήσουμε μια τέτοια μέθοδο η οποία θα διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη επιδιώκουν τους σωστούς στόχους, τους υιοθετούν, τους κάνουν ιδιοκτησία τους και τους επιδιώκουν βεβαίως με νόμιμα μέσα. Και μια ε, συμπληρωματική ερώτηση. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε κύριε Επίτροπε, την ερώτησή μου δεν την απαντήσατε συγκεκριμένα. Και εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν επενδύσει, παιδεία, οικολογική οικονομία. τι όμω το εξή ερώτημα. Πώ μπορούμε να εμποδίσουμε ένα τμήμα, ένα αριθμό των κρατών μελών να μας ε, αναχαιτίζει με λανθασμένη φορολογική πολιτική, ε, με λάθο χρήση της ε, κατανάλωση και με τον τρόπο αυτό καταλήγουμε στο να υπάρχουν αυξημένε δαπάνε σε ορισμένα κρατημέλη και χαμηλότερε σε άλλα. Υπάρχει λοιπόν μια ανισορροπία στην Ευρώπη η οποία θέτει σε κίνδυνο την οικονομία τη και θέλω να ακούσω πιο συγκεκριμένα τι προτίθεστε να κάνετε για να επικρατήσει μια ισορροπία στην οικονομία των κρατών μελών. Είναι αλήθεια ότι γίνεται ευρύτατα λόγος για τις ε, παγκόσμιες ε, μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες η Ευρωπαϊκή, Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν και εκείνες λόγο για πλεονάσματα και λύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι είναι πιο ισορροπημένη και έχει μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Βεβαίως πολλά, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν, ε, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους. Η, το όλο θέμα που ε, θέτεται επιτάπητος ε, έχει μεγάλη σημασία, έχει σχέση με την μακροοικονομική ισορροπία και εγώ αν καταλάβω τη θέση του Επιτρόπου, προτίθεμαι τη συζήτηση αυτή να την οδηγήσω σε βάθος, σε ενδελεχή ανάλυση. Να δούμε ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν στην ανισορροπία και να δούμε βεβαίως κατά πόσον ενδεχομένως αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξή της ε, και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Καταλήγω να σας πω, επιτρέψτε μου, έχω ανοιχτό και φρέσκο μυαλό. Ο κύριος Έπιν. Ευχαριστώ. Και καλωσορίζω εδώ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν δούμε την Ευρωζώνη, φαίνεται ένας πολύ ωραίος ε, καθρέφτης που χωρίζεται όμως στη μέση. Ε, βλέπουμε ότι έχουν ξεφύγει κάθε ελέγχου τα δημόσια οικονομικά. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν να συμμορφωθούν στα κριτήρια της, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι έχετε τις δυνατότητες, το χαρακτήρα, τη πυγμή να σταθείτε απέναντι σε μεγάλες πολλές φορές χώρες μέλη που δεν τηρούν τα κριτήρια ε, που έχουμε βάλει για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και όταν υπάρχουν χώρε οι οποίε επιμονή μου βάσης ε, δεν ε, τηρούν τα κριτήρια και κάνουν κατάχρηση τη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ένωση, τι θα κάνετε γι' αυτά. Thank you for this, uh, this question. Uh, I leave the question of my... Ρωτάτε κατά πόσο είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω με πυγμή αυτές τις υποθέσεις. Κοιτάξτε, έχω κάποιο υπόβαθρο. Ήμουνα και αρμόδιος επίτροπος για τις διαπραγματεύσεις για τις εντάξεις νέων χωνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οπότε, όταν ε, μιλάμε για αυτά τα θέματα, μερικές φορές λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχει. Μερικές φορές χρειάζεται πειθό, χρειάζεται περισσότερο πειθό. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν, παίρνουν τελικά τις αποφάσεις, τις τελικές για κάθε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η κάθε απόφαση κλειδί απαιτεί ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Από τη θέση αυτή, πάντως, έχω περισσότερες αρμοδιότητες χάρη στο Σύμφωνο Σταθερότητας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εφόσον χρειαστεί θα χρησιμοποιήσω όλες τις δυνατότητες που ε, μου δίνουν τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου για να διασφαλίσω ότι τα μέλη της ε, Νομισματικής Ένωσης θα κάνουν αυτά που πρέπει. Για να είμαι συγκεκριμένο για την Ελλάδα, για παράδειγμα, αν τελικά δεν ελεγχθούν τα δημόσια οικονομικά της, θεωρείτε ότι είναι δυνατότητα να εγκαταλείψει την ε, Ευρωζώνη. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Όχι, δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει ότι πολύ σοβαρά θα φροντίσει να λύσει το πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με ανησυχίες βέβαια την υπόθεση. Είχαμε μια τεχνική αποστολή στην Ελλάδα και αυτό το μήνα, τον επόμενο, θα αντιμετωπίσουμε την υπόθεση της Ελλάδας και το θέμα του υπερβολικού ελλείμματος. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα πάρουμε αποφάσεις, θα κάνουμε συστάσεις και εννοείται ότι συνεργαζόμαστε με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι Εσωτική σημασία σε ελληνική κυβέρνηση σύντομα μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να μην πω μέρες θα παρουσιάσει ένα συνολικό πακέτο πολιτικής με συγκεκριμένα και απτά μέτρα προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα που είναι της τάξης του 12 με 13%. Ευχαριστώ. πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρεν, στην εισαγωγή σας ε, τοποθετηθήκατε αδιαμφισβήτητα στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και σε αυτήν επανέρχομαι και εγώ. Αν σας κατάλαβα καλά, η κοινωνική οικονομία της αγοράς σημαίνει ότι το κράτος διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία και επίσης σημαίνει ότι το κράτος ε, είναι και ενεργός παράγων στην αγορά εργασία. Στις σκανδιναβικέ χώρες αυτό σημαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τον τρόπο αυτό οι σκανδιναβικέ χώρες τα τελευταία 10-15 χρόνια κατόρθωσαν να μειώσουν σημαντικά την ανεργία. Εσείς λοιπόν έρχεστε από τη Φινλανδία και γι' αυτό σας ερωτώ όσον αφορά αυτό το ρόλο του κράτου ε, ω ε, οικονομικού παράγοντα και εργοδότη αν θέλετε, ε, ποια είναι η δική σα άποψη. Ε, και θεωρείται ότι αυτός ο ρόλος του κράτους ε, πρέπει να ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω και μήπως έχετε μιλήσει με την Ισπανία και η Ισπανία συμφωνεί άραγε μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Κλούιτο. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εγώ είμαι πεπισμένος ε, για την ορθότητα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Γιατί είναι αποτελεσματική και γιατί είναι εκείνη η οποία προσέφερε αυτό το ευρωπαϊκό ε, μοντέλο κοινωνίας το οποίο συνδυάζει αφενός τον επιχειρηματικό δυναμισμό και αφετέρου την κοινωνική αλληλεγγύη. Για μένα λοιπόν το κράτος ε, πράγματι καλείται εδώ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Όταν παραδείγματο χάρη μιλάμε για τη στρατηγική του 2020 ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο θα δύναται και θα ε, πράξει τελικά την οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις καινοτομίες, μέσα από την πράσινη οικονομία, τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες και θα βελτιώσει τόσο το δημόσιο όσο προφανώς και τον ιδιωτικό εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το κράτος και η αγορά μπορούν να συνεπάρξουν. Καθοριστική σημασία είναι το να αναζητηθεί η κρίσιμη ισορροπία, γιατί το κράτος είναι εκείνο που ευθύνεται για τον καθορισμό των πλαισίων, για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Συμπληρωματική ερώτηση. Ένα ε, σημαντικό σημείο είναι ο ρόλος ε, του κράτους ε, ως οικονομικός παράγων στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Και οι ιδιωτικοποιήσεις ε, δρομολογούνται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ στη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εσάς. Εσείς τι ακριβώς πιστεύετε για την πολιτική ιδιωτικοποίησεων. οι ιδιωτικοποιήσει αυτές καθεαυτές δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν λελογισμένα από τα κράτη-μέλη και εναπόκειται στα ίδια τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πώς ακριβώς επιθυμούν να διοργανώσουν τόσο το δημόσιο τομέα όσο και τα κοινωνικά τους. Η Κομισιόν λοιπόν προτίθεται να καταθέσει μια πρόταση, ένα πλαίσιο ποιοτικό για τις ε, δημόσιες ε, υπηρεσίες και τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και εγώ από δική μου πλευρά θα συμβάλλω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής οικονομίας αγορά. Το να έχουμε δηλαδή ε, έναν εύρυθμα λειτουργούντα δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα που να είναι αποτελεσματική. Ο κύριος Μπλουμ. Ο κύριος Μάρτιν από τους ανεξάρτητους. Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά την ε, διαδικασία, μας είπατε, απαντώντας την ερώτηση 3, ότι επιθυμείτε να διασφαλίσετε την πρόσβαση στην ε, ενημέρωση, όπως το είχα ζητήσει και εγώ ως Ευρωβουλευτής, νομίζω και εσείς. Τότε το λόγος ε, για ε, τη διαφάνεια και για το Lobbying Act που συζητείται τότε στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Ερωτώ λοιπόν, οι αρχές που ε, καθορίζουν αυτή τη διαφάνεια είναι σημαντικές για σας, θα τις προβάλλετε και με ποιον ακριβώς τρόπο εξοπλίζεστε στο να αντιμετωπίσετε αυτές τις τεράστιες πιέσεις που θα ασκηθούν από τις ομάδες πίεσης και πώς θα τα ανακοινώνετε και θα τα γνωστοποιείτε όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εγώ ξέρετε έχω κατά νου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις ομάδες εργασίας. Πιο συγκεκριμένα αναφερθήκατε σε όλα αυτά περί διαφάνειας και των, της νομοθεσίας. Τι ακριβώς Πώς εννοείται με αυτά. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν για αυτήν την ερώτηση. Πράγματι, πριν από πολύ καιρό, πριν από δέκα χρόνια, ε, ήμουνα τότε στην Επιτροπή και τότε καταρτίζαμε τον κώδικα συμπεριφοράς και τους κανόνες της διαφάνειας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο προϊόν και είμαι δεσμευμένος απέναντι σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι και δικό μου όσον αφορά αυτόν τον κώδικα συμπεριφορά. Είναι πολύ πιο σύγχρονο το εργαλείο αυτό, αν το συγκρίνει κανεί με τον κώδικα συμπεριφορά για τη διαφάνεια του κράτου των κρατών μελών που γνωρίζω καλύτερα, των σκανδιναβικών. Στη Φιλανδία, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν 34 εξαιρέσει στη διαφάνεια και ε, συχνά γίνεται χρήση αυτών. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε πολύ λιγότερες εξαιρέσεις και είμαστε πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά τους κανόνες περί διαφάνειας. Εγώ λοιπόν θα συνεργαστώ με τον ε, πρόεδρο κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Σεύκο που ε, θα είναι αρμόδιος εφόσον ε, αναλάβει αυτό το αξίωμα και θα με έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και το βέλτιστο κώδικα συμπεριφοράς σε σχέση με τις ομάδες πίεσης. Εγώ θέλω να σας πω, θεωρώ και βασίζομαι στο ότι όλοι οι κοινοτικοί θεσμοί θα βασιστούν στο μέλλον ε, σε αυτόν τον κώδικα συμπεριφορά. Δεν πρέπει να ανησυχείτε για μένα, ούτε εγώ για εσά όσον αφορά τι ομάδε πίεση. Για να είμαι ειλικρινή, εγώ προτιμώ να φάω το βράδυ με την οικογένειά μου από το να βρεθώ σε ένα επίσημο δείπνα, δείπνο με ε, κάποια ομάδα πίεση. Χωρί βέβαια να θέλω να προσβάλλω κανένα. Έχετε και άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Ε, δεν συμφωνούμε μόνο σε αυτό, από ό,τι φαίνεται και σε πολλά άλλα. Παρ' όλα αυτά, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμένη στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Η καγκελάριος του μεγαλύτερου κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ένα στόχο όπου όλοι οι παράγοντες, όλα τα προϊόντα και όλες οι περιοχές θα υπάγονται σε έλεγχο. Αναφέρομαι κυρίως στη χρημα, στις χρηματοψηφιτικές αγορές. Δεν ξέρω αν είσαστε αρμόδιος για τις χρηματοψηφιτικές αγορές, αλλά εσείς μιλάτε και με το πνεύμα της αλληλεγγύης. Προτίθεστε λοιπόν στην Επιτροπή να προωθήσετε αυτό το θέμα του ελέγχου των χρηματοψηφιτικών αγορών ή όχι. Και πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την νομοθεσία περί διαφάνειας ε, προτίθεστε αυτή να την ε, εφαρμόσετε και στο δικό σας τον τομέα αρμοδιοτήτων. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε πάρα πολύ γρήγορα και συντομότατα. Με δύο απλά ναι. Κοιτάξτε, ξεκινάω με το τελευταίο. Εγώ βεβαίως και είμαι φύλλα διακείμενος ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετώ άκρητα τα μοντέλα των Ηνωμένων Δεύτερον, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, όσον αφορά την εποπτεία σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο κύριος Μπαρνιέ, ο ε, προτινόμενος επίτροπος, θα είναι αρμόδιος για ε, χρηματοψηφιακούς ε, κανονισμούς σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Θα συνεργαστούμε. Εγώ συμμετείχα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε προτάσεις για το πακέτο που έχει κατατεθεί σχετικά με την εποπτεία σε μάκρο και μικροοικονομικό επίπεδο. Εμένα με αφορά περισσότερο το μικρο επίπεδο, η μικροοικονομία. Πρόκειται να είμαι ε, μέλος ε, του Συστημικού Συμβουλίου, ε, το οποίο θα ασχοληθεί με αυτό το πακέτο, όπως σας είπα και προηγουμένως. Έφτασε ο κύριος Μπλουμ. Έχετε ένα λεπτό. Σα Thank you very Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη μου άφηξη. Είμαι τυχερός που έφτασα. Καθυστερημένα σας λέω καλή χρονιά κύριε Ρέν. Έχω μια σοβαρή ανησυχία ότι οι πολιτικοί άντρες δεν έχουν μάθει πολλά από τις πρόσφατες κρίσεις και αποτυχίες που είχαμε. Πρέπει να πούμε ότι η αρχή αυτής της κρίσης ήταν στη δεκαετία του 70 με την νομοθεσία για την επανεπένδυση, το οποίο δεν είναι και πολύ καλός νόμος. Τον ε, ε, υπέβαλε ο πρόεδρος Κάτερ και μείωσε τις απαιτήσεις προσοχής που είχαν οι τράπεζες. Αυτό οδήγησε σε λιγότερη εποπτεία από τις κεντρικές τράπεζες και αυτό το ίδιο συνέβησε, συνέβη μετά σε όλα τα βιομηχανικά κράτη με εξαίρεση την Αυστραλία-Ασία. Μερικοί επόπτες οι οποίοι ακόμα υπάρχουν δεν έκαναν σωστά την εποπτεία τους. Ε, ένα λεπτό μόνο για το ερώτημά σας είχατε, λέει η Πρόεδρος και ακόμα δεν έχετε θέσει ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι θα διδαχθούμε από τις εμπειρίες που είχαμε προηγουμένως και θα ασχοληθούμε όπως πρέπει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τους ε, τραπεζίτες και τους, τις κεντρικές τράπεζες. Ο κύριος Ρεν. Κατανοώ ότι θέτεται ένα ερώτημα για το πακέτο που αφορά τον τραπεζικό τομέα και την εποπτεία του και σχετίζεται με τα διδάγματα. Κατά την άποψή μου, καλό θα ήταν οι συνομοθέτες, το, το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, να μπορέσουν να υιοθετήσουν αρκετά σύντομα το νομοθετικό πακέτο για την μακροοικονομική εποπτεία. Γιατί μας χρειάζεται επιγόντως και κατά την άποψή μου είναι ένα θετικό βήμα για να εξασφαλίσουμε ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός και η εποπτεία θα λειτουργήσουν σωστά στην Ευρώπη και ελπίζουμε και παγκοσμίω. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Εκπροσωπούσα πριν μερικές εβδομάδες την Κομισιόν στο Συμβούλιο όταν είπα ξεκάθαρα και τους μίλησα ως Επίτροπος για θέματα διεύρυνσης, αντικαθιστώντας την κυρία Βάλστρομ και τους είπα ότι θα θέλαμε πιο δεσμευτικές εξουσίες στον τομέα των δημοσιονομικών, οικονομικών και προληπτικής μακροοικονομικής εποπτείας και ελπίζω να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο ώστε να έχουμε επαρκή εποπτεία στο τέλος. έχετε 20 δευτερόλεπτα για μια συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τελικά η, η εσφαλμένη νομοθεσία της δεκαετίας του 70 μας οδήγησε σε όλα αυτά. Θα, απάντηση. Θα κοιτάξω τα ιστορικά βιβλία για να βγάλω τα διδάγματα από αυτή την νομοθεσία. Πάντως κατάλαβα το επιχείρημά σας Υπάρχει μεγάλη ιστορία τέτοιου είδους προκλήσεων στις κοινωνίες μας. Τώρα οι επίγουσες προκλήσεις είναι να αντιμετωπίσουμε τη δημοσιονομική κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να υιοθετήσουμε αυτό το πακέτο από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ομαδικές ερωτήσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά μία κάθε φορά ερώτηση. Ο κύριος Λάγκεν πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εσείς αναλάβατε έναν από τους δυσκολότερους τομείς, ε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ε, κατ' ουσίαν έχει ακυρωθεί γιατί τα ε, επιτόκια παρουσιάζουν μεγάλε αποκλήσει, ορισμένε χώρε βρίσκονται στα πρόθυρα τη χρεοκοπία και μετά από ερώτηση απαντήσατε ότι θα αναζητήσετε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να δρομολογήσετε τη σταθερότητα. Εγώ θέλω να σα πω ότι αυτό δεν αρχική. Τα κράτη είναι εκείνα που θα πρέπει να προβούν σε μεταρρυθμίσει ε, και να ξεπληρώσουν τα χρέη του. Και δεν μπορούν να θεωρούν ότι η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας ερωτώ, πώς τα φαντάζεστε όλα αυτά. Τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα, ποια είναι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να δρομολογηθούν μεταρρυθμίσεις και πράγματι ο δανεισμός και το εξωτερικό χρέος να μειωθούν ρίζικα, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά τέτοιους καταστάσεις αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τη σταθερότητα του ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ερώτηση, ε, κύριε Λάγκεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον του ευρώ και να ενισχύσουμε την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Εδώ λοιπόν το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας μας προσφέρει το πλαίσιο για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε υγιή δημόσια οικονομικά. Ε, σε αυτό το πλαίσιο οι στρατηγικές εξόδου είναι καθοριστική σημασίας. Πρέπει να εφαρμοστούν σωστά. Πρέπει να υπάρχει σωστός συντονισμός και να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ιδιαιτερότητα των κρατών μελών. Να υπάρχει μια ε, σωστή αλληλουχία μέτρων που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής εξόδου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε και συμφωνεί εδώ η Επιτροπή και εγώ προσωπικά συμφωνώ ότι η φορολογική σταθεροποίηση θα πρέπει να αρχίσει το λιγότερο το 2011. Σε ορισμένες χώρες ίσως και νωρίτερα, καθότι έχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα και έχουν περιορισμένο χώρο κινήσεων φορολογικών. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, όλα αυτά μπορούν να συμβούν μόνο εφόσον έχει δρομολογηθεί, έχουν δρομολογηθεί οι μεταρρυθμίσεις. Το 1937 είχαμε κάνει την εμπειρία, το 1990 στην Ιαπωνία επίσης. Πρέπει λοιπόν να ε, είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και από τη στιγμή που οι οικονομίες βασίζονται σε υγιή θεμέλια, τότε θα κληθούμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Συμπληρωματική ερώτηση. Αναγνωρίζουμε ότι ήσασταν πολύ αποτελεσματικός ε, ως ε, αρμόδιος για τη διεύνηση. Δεν συμφωνήσαμε πάντα. Εσείς ε, προβάλλατε και φέρατε τη διεύνηση παρότι φέρατε και πάρα πολλά προβλήματα. Και τώρα τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξετε τη στρατηγική. Τώρα πρέπει να δείξετε θάρρος γιατί αλλιώς κινδυνεύει το ευρώ. Την δική σας την πολιτική θα μπορέσετε να την εφαρμόσετε αν κρυθεί απαραίτητο και ενάντια στον κύριο Αλμούνια. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον ε, συνάδελφο και φίλο μου Γιωακή Μαλμούνια. Και μάλιστα ε, προτίθεμαι σε πάρα πολλές περιπτώσεις να μελετήσω αυτά που έχει επιτύχει και να ακολουθήσω και τα ίχνη του, αν αυτό είναι δυνατόν. Στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι καθοριστική σημασίας και βεβαίως Παράλληλα υπάρχει και το Σύμφωνο Σταθερότητας το οποίο προσφέρει τα νομικά εκείνα εργαλεία που επιτρέπουν να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν τους κανόνες που έχουν κριθεί από εμά στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θέλω να σας πω το εξής. Ε, σύντομα θα γίνει η δοκιμή, το τεστ, αν όλα βαίνουν καλώς. Γιατί πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσουμε μια κρίσιμη κατάσταση με την Ελλάδα, είτε στο τέλος αυτού του μήνα, είτε στις αρχές του επόμενου. Εκεί θα ληφθεί η απόφαση σε σχέση με το υπερβολικό έλλειμμα και τότε θα κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Επόμενο ερώτημα σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τις προτεραιότητάς σας. Η... Τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά είναι ένα από τους τρεις. Είναι προφανές αυτό. Γιατί είναι ένας από τους μηχανισμούς, ένα από τα εργαλεία της Ένωσης. Αλλάξαμε πριν μερικά χρόνια το Σύμφωνο Σταθερότητας και το κάναμε πιο ευέλικτο και αυτό το χρησιμοποίησαν πολλά κράτη-μέλη και τελικά μπήκαμε στην κρίση και ένας μεγάλος αριθμός κρατών μελών είχαν χρησιμοποιήσει ήδη τα όσα επέτρεπαν οι κανόνες και δεν είχαν την δυνατότητα να αντιδράσουν όταν έφτασε η κρίση και είδαμε ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα. Πώς θα ενισχύσετε το σύμφωνο σταθερότητας. Ίσως με την ιδέα να υπάρχουν πλεονάσματα τους, τις καλές εποχές αλλά αυτό θα μπορέσει να μας κάνει να σεβαστούμε τους κανόνες τους δύσκολους καιρούς. Είστε διατεθειμένος να προτείνετε κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μας, κατά την άποψή μου, η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη μας έδωσε αρκετά καλά αποτελέσματα και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης. Τα κράτη-μέλη μας μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιπλέον ευελιξία έδωσε αυτή η μεταρρύθμιση σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά την άποψή μου, το άτος 2009 και το 2010 αντιμετωπίζουμε εξαιρετικές περιπτώσεις τώρα που έχουμε οικονομική κρίση και ύφεση. Αυτό σχετίζεται μάλιστα και με ένα προηγούμενο ερώτημα. Δεν είχα προηγουμένω το χρόνο να εξηγήσω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυστηρότητα στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και με αυτή τη λογική πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ευρύτερη εποπτεία συμπεριλαμβανομένων και εποπτείας για μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εισαγάγουμε μεθόδους εις βάθους εποπτείας με βάση τη νέα συνθήκη η οποία στο άρθρο 121 και 136 δίνει τέτοιου είδους δυνατότητες. Σκοπεύω να παρουσιάσω μια ανακοίνωση για ενισχυσμένο συντονισμό οικονομικών πολιτικών και εποπτεία στην αρχή της θητείας μου, μόλις αναλάβω τα καθήκοντά μου εάν εγκριθώ και αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και τους καλούς καιρούς όπως είπατε. Συμπληρωματικό ερώτημα. Να είμαι πιο συγκεκριμένος. Είστε διατεθειμένος να συζητήσετε ή να προτείνετε αυστηρότερες απαιτήσεις για τα πλεονάσματα τους καλούς καιρούς, διότι αν τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο να έχουν ελλείμματα στις καλές εποχές, στην ουσία δεν θα μπορούν να σεβαστούν τους κανόνες τις δύσκολες εποχές, όποια και αν είναι η ευελιξία. Αυτό θα είναι, μπορούσε να είναι ένα από τα βασικά διδάγματα από αυτήν την κρίση. Απάντηση. Το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι στην καρδιά των συζητήσεων για την ενίσχυση της εποπτείας των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε δίκιο. Οι χώρες οι οποίες μπήκαν στην οικονομική κρίση με σχετικά υγιή δημόσια οικονομικά είχαν αρκετό φορολογικό περιθώριο για να δώσουν κίνητρα αντικυκλικά κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Οπότε υπάρχουν επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτή τη λογική ενστικτοδός θα πήγαινα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά καλύτερα είναι να τα αναλύσουμε όλα αυτά εις βάθος και θα ήθελα να επανέλθω με μια πιο εις βάθος πρόταση εάν με εγκρίνεται στα καθήκοντά μου. Κύριος Τίσεν. Ε, Η κυρία Τίσεν. Κύριε Πίτροπε, άμα θέλετε την κοινωνική οικονομία, πρέπει να ακολουθήσετε τους στόχους της συνθήκης. Μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, αλλά περισσότερη πράσινη ανάπτυξη με περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πολλοί από εμά εδώ προσδοκούμε από την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, όμως αυτό που φοβούνται πολλοί συνάδελφοι εδώ είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αρκετά ώστε να πετύχουμε το στόχο μας και να είμαστε αποτελεσματικοί. Εσείς είπατε πριν και το έχω σημειώσει ότι οι μηχανισμοί εποπτείας του Συμφώνου Σταθερότητας θα δώσουν νέα πνοή στη νέα στρατηγική. Ναι, αλλά τελικά το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό. Ξέρουμε ότι το naming and shaming δεν έχει δουλέψει αρκετά, το να κατονομάζουμε τους φταίχτες. Γιατί όμως. Και τι άλλο προτείνετε εσείς. Δεν λέω να δουλεύουμε με κυρώσεις, αλλά τουλάχιστον να δίνουμε έναν έπαινο με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάτι υπέρ του καλού μαθητή στην τάξη. Συμφωνώ για το ότι πρέπει να μελετήσουμε την εμπειρία που είχαμε μέχρι τώρα από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες, αλλά υπήρξαν και κάποιες επιτυχίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια πιο κοινή άποψη μεταξύ μας όσον αφορά την αγορά εργασίας. Με την ευελιξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας, με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, είδαμε τι κάνανε γι' αυτό. Συγχρόνως υπάρχουν και αδυναμίες στη στρατηγική της Λισαβόνας όπως είπαμε. Εντοπίζονται η μία είναι ότι δεν είχαμε αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου εποπτείας και δεύτερον δεν υπογραμμίζαμε αρκετά τις δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία μπορούν και πρέπει να διορθωθούν. Για το πρώτο, δεν βλέπω εγώ τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο να βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε εταίροι μεταξύ μας όλοι και αν θέλουμε η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 να πετύχει, φυσικά και χρειαζόμαστε τα κρατη τα συνδικάτα και όλους τους υπόλοιπους ε, εταίρους να ε, συμμετέχουν και να δρουν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και οικονομική ε, ανάπτυξη και για θέσεις εργασίας, για την απασχόληση. Από την άλλη μεριά, χάρη στην εταιρική σχέση μεταξύ μας, μπορέσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο για την επίτευξη κοινών στόχων. Σίγουρα αυτό θα είναι στην καρδιά από εδώ και πέρα. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, μια μικρή ακόμα ερώτηση κύριε Επίτροπε. Θέλω να ξέρω κατά πόσο είσαστε έτοιμος να ερευνήσετε τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη που κάνουν προσπάθειες να ανταμείβονται με κάποιο τρόπο. Και τα κράτη-μέλη που δεν κάνουν καμία προσπάθεια για να πετύχουν τους στόχους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να έχουν κυρώσει σε βάρος τους. Είσαστε διατεθειμένος για κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού και των αποφάσεων για τη στρατηγική Ευρώπη του 2020 πρέπει να δούμε και τα κίνητρα και τα μέσα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχει η στρατηγική μας αυτή. Πιθανόν λοιπόν να εξετάσουμε και εγώ είμαι έτοιμος να εξετάσω κίνητρα υπέρ των κρατών μελών για να πετύχει η στρατηγική μας αυτή. Είπα και στην αρχή, στην εισαγωγή μου, ότι θέλω αξιολόγηση των μηχανισμών που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε μετά τι νέες προτάσεις μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη απόδοση των χρημάτων που ξοδεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλδημοκράτες τώρα ερωτήσεις. Η Πέρανς Πέρες έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπο, έχετε ένα πολύ θεμελιώδες χαρτοφυλάκιο, απαιτεί φαντασία, αντιμετωπίζει προβλήματα το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά και πριν την κρίση δεν μας επέτρεψε να έχουμε σύγκληση των οικονομιών ακόμα και στην Ευρωζώνη. Και αυτό που απέδειξε αυτή η κρίση είναι ότι υποφέρουμε από την όλο και μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές οικονομίες, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αντέξει η Οικονομική Ένωση. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να διορθώσετε αυτή την κατάσταση. Μιλήσατε για καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Μήπως τώρα πρέπει να θέσουμε το θέμα για κοινή διαχείριση του χρέους, την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων πέρα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό ως αντάλλαγμα των νέων εργαλείων εποπτείας. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε προηγούμενες μου απαντήσεις για να γλιτώσουμε χρόνο σε ό,τι αφορά το συντονισμό και την εποπτεία των δημοσιονέμων οικονομικών. Συμφωνώ μαζί σας ότι από την κρίση μάθαμε το δίδαγμα ότι θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας και αυτό θα είναι ένα από τα βασικά μελήματα της επόμενης Επιτροπής μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο. Αναφερθήκατε στα νέα εργαλεία χρηματοδότησης, ευρωπαϊκά ομόλογα ή άλλου είδους ευρωπαϊκά ομόλογα. Κατά την άποψή μου, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση παραδείγματο χάρη υποδομών, τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αξιολογηθεί εις βάθος και έχω ανοιχτή θέση σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση τέτοιου είδους προγραμμάτων μαζί και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραδείγματο χάρη. Ήδη με κάποια λογική υπάρχουν ήδη τέτοιου είδους μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει εγγυήσει για τέτοιου είδους επενδύσεις, τέτοιου είδους προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξεταστεί το θέμα και έχω ανοιχτή θέση για το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι όλες οι δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να έχουμε δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης για να επιτύχουμε τους στόχους του προγράμματος 2020 για οικονομική μεγένθηση και αύξηση της απασχόλησης. Σας ευχαριστώ. Με αυτή τη λογική, τι πιστεύετε για την πρωτοβουλία που επιτρέπει να θέσουμε το οικονομικό ερώτημα στα πλαίσια της γεωπολιτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλάω εδώ για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεκάλεσε ο Ευρωπαϊκός Πρόεδρος Βαν Ρομπέ για την 11 Φεβρουαρίου και νομίζετε ότι μπορούμε να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και να το επιτύχουμε αυτό χωρίς να μπορείτε να υποπτεύετε στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου σας τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Απάντηση. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε στενά και αποτελεσματικά με τον συνάδελφό μου προτινόμενο επίτροπο κύριο Μισελ Μπάρνιε σε ό,τι αφορά την μικρο και μακροοικονομική εποπτεία και το σχετικό κανονισμό. Ήδη έχουμε συζητήσει το θέμα μαζί και θα συνεχίσουμε να το συζητούμε με την προϋπόθεση βεβαίως ότι και οι δύο θα εγκριθούμε ως Επίτροποι. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέλει να κατευθύνει αυτό το ίδιο ισχυρά και την στρατηγική για το 2020. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μπαρόζο, ο ίδιος ανέλαβε τα ενία αυτής της προσπάθειας. Ο ρόλος μου θα είναι να τον βοηθήσω στα πλαίσια του συντονισμού οικονομικών πολιτικών για οριζόντια θέματα και έχω την πρόθεση να κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δεσμευτεί για αυτήν τον συντονισμό οικονομικών πολιτικών που συζητήσαμε προηγουμένως. Εγώ βεβαίως δεν θα είμαι παρόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα είναι παρόν ο Πρόεδρος Μπαρόζο. Αλλά έχουμε την ίδια άποψη για το θέμα. Επόμενο ερώτημα. Κύριε Επίτροπε, προηγουμένως αναφερθήκατε σε κάποια επιστροφή σε υγιή δημοσιονομικά για την στρατηγική εξόδου. Όμως το 2010 θα έχουμε μέγενθος ανάπτυξη μικρότερη του 1%. Μήπως είναι πρόωρο να επανέλθουμε σε πολύ αυστηρά δημόσια οικονομικά γιατί αυτό θα είναι εις βάρος της ανάπτυξης. Και αν χρειαστεί να διατηρηθούν όλα αυτά τα μέτρα στήριξης. Η αποτελεσματικότητα κάθε δημόσιας επένδυσης θα πρέπει να αξιολογηθεί, διότι δεν θέλουμε κάποια αμφιλεγόμενα φορολογικά μέτρα να καταδικάσουν τις πολιτικές αυτές. Κύριε Επίτροπε, θα κάνετε μελέτη εφικτότητας σε ό,τι αφορά τα φορολογικά μέτρα που μαζικά έχουν λάβει κάποιες χώρες. Uh, uh, Έχετε δίκιο η Ευρώπη υποφέρει από πρόβλημα ανάπτυξης και το δυναμικό της ανάπτυξής μας αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται στο έπακρο. Θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουμε στην βέλτιστη χρήση των δυνατοτήτων μας για ανάπτυξη. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να συνδυάσουμε δύο πράγματα και αυτό σχετίζεται με το πρώτο τμήμα του ερωτήματός σας. Πρέπει να συνδυάσουμε επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές στην παιδεία, στην καινοτομία, σε περιβαλλοντικές, ενεργειακές τεχνολογίες και ταυτόχρονα πρέπει να αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι στρατηγικές εξόδου από την κρίση, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Η πρώτη καμπύλη λοιπόν πάει προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τις ανάγκες επενδύσεων. Η δεύτερη πάει προς τα κάτω ή τουλάχιστον είναι σταθερή. Του του εάν δεν διορθώσουμε την τάση των δημοσίων μας οικονομικών, θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου απλώς θα χρηματοδοτούμε το χρέος μας. Θα χρησιμοποιούμε όλους τους πόρους μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους και δεν θα μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις. Πρέπει να βρούμε τη σωστή οδό και πρέπει να δημιουργήσουμε καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης και να συνδυάσουμε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Συμπληρωματικό ερώτημα. Στα πλαίσια των πολιτικών εξόδου πρέπει εξ ονόματος της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών να μειώσουμε τις συντάξεις και τις κοινωνικές δαπάνες ενώ αυτές οι δαπάνες έχουν αντικυκλικό αποτέλεσμα όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Απάντηση. Συμμερίζομαι την άποψή σας ότι στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο οι δημόσιες και οι κοινωνικές υπηρεσίες μεταξύ των οποίων είναι και οι υπηρεσίες υγείας διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Όμως για να έχουμε βιώσιμο κράτος χρειάζονται βιώσιμα δημόσια οικονομικά θα πρέπει τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων, γιατί μιλάμε εδώ για εθνικές αρμοδιότητες, στην κατανομή του προϋπολογισμού τους, τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν ποιες είναι οι προτεραιότητες τους χρηματοδότησης. Είναι απαραίτητο κατά την άποψή μου τα κράτη-μέλη στους προϋπολογισμούς τους να βελτιώσουν την ποιότητα των δημοσίων τους οικονομικών και να έχουν στόχους που θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν μια πιο έξυπνη και πράσινη οικονομία. On Εκ μέρους λοιπόν των φιλελευθέρων ο κύριος ε, Κλίντς. Κύριε Ρέν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, τονίζουν ε, επανειλημμένα το πόσο πολλοί επιθυμούν να συνεργαστούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση από κοινού και να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθεί μια παρόμοια κρίση. Εγώ λοιπόν έχω την εντύπωση, πρέπει να σας πω, ότι η πραγματικότητα είναι τελείως αντίθετη. Δηλαδή ότι υπάρχει πλήρης απόκληση. Σκεφτείτε την ε, κεφαλαιοποίηση των ε, τραπεζών, τα λογιστικά, τον τρόπο υπολογισμού λογιστικών ε, έχω λοιπόν την εντύπωση ότι σήμερα η Ευρώπη είναι πολύ πιο μακριά από την Ευρώπη από ό,τι αν θέλετε πριν από τρία χρόνια. Η ερώτηση λοιπόν που σας υποβάλλω είναι πολύ συγκεκριμένη. Τους επόμενους 12 μήνες τι προτίθεστε να κάνετε πολύ συγκεκριμένα για να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει ε, ο πειρασμός ε, να ξαναγίνει χρήση του περίφημου αρμπιτράζ. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς. Συμφωνώ εν μέρη με αυτά που είπατε και εν μέρη διαφωνώ προφανώς. Συμφωνώ μαζί σας ότι πράγματι πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Και παράλληλα, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, κυρίως στο πλαίσιο της ομάδας των G20, συμφωνήσαμε και οι δυο μας ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει ένα πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν το 2008 και είχαν ως στόχο να αποφευθεί η τρέχουσα ύφεση, να εξελιχθεί σε μία ε, ύφεση μακράς διαρκείας, σε ένα κράχ. Όσον αφορά τη νομοθεσία, αναφέρθηκε σε αυτήν, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανονισμούς και στην εποπτεία. Πράγματι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και έχω κατά νου κυρίως ε, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η Κίνα είναι μια οικονομία πλεονασματική η οποία δεν είναι πρόθυμη να δεχθεί υποτίμηση του νομίσματός της. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ελληματική οικονομία με μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε σοβαρές συζητήσεις με τους βασικούς μας εταίρους, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα, για να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ισορροπία σε παγκόσμιο μακροοικονομικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν η Κίνα είναι εξίσου σημαντική όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν μιλάμε για μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κύριε Ρέν, μία συμπληρωματική ερώτηση στην Ευρωζώνη και στη διεύρυνσή της. Υπάρχουν οικονομολόγοι που ισχυρίζονται ότι θα ήταν σκόπιμο τα νέα κράτη-μέλη των οποίων ε, το νόμισμα συνδέεται έτσι και το ευρώ, όπως η Λετωνία, να ενταχθούν στην Ευρωζώνη το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα τους προσέφερε ασφάλεια και θα εξάλληφε τον κίνδυνο ότι θα μπορούσε να υποτιμηθεί το νόμισμά τους. Εσείς ε, τι πιστεύετε γι' αυτό το ενδεχόμενο μιας ε, ταχύτατης, σύντομης ένταξης της οικονομίας αυτών των χωρών στην Ευρωζώνη. Κατά τη δική μου άποψη πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες και τον νόμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα ε, νόμων και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία της. Γνωρίζω πολύ καλά τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους και δικηγόρους. Το λέω απλά όσον αφορά την ερμηνεία της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι σαφές ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι να υπάρχουν υγιή, μακροπρόθεσμα, δημοσιονομικά, μακροοικονομική σταθερότητα τα πέντε κριτήρια σύγκλησης είναι δείκτες που μας επιτρέπουν να μετρήσουμε το κατά πόσον μια χώρα καλύπτει αυτά τα εκ των όνου κριτήρια για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά τους, ε, το ενδεχόμενο των υποψηφίων, θα πρέπει βέβαια να ερευνήσω για να δω κατά πόσον οι χώρες αυτές ε, εφαρμόζουν και σέβονται τους κανόνες και τον νόμο της νομισματικής ένωσης. Ε, κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για κανόνες, οι συμπληρωματικές ερωτήσεις δεν θα πρέπει να αφορούν τελείω διαφορετικό θέμα, να είναι επί του ιδίου θέματο. Γι' αυτό λοιπόν σα παρακαλώ να μην ακολουθήσετε το παράδειγμα του κυρίου Κλίντ. Κοιτάξτε, η Φιλανδία με έχει συνηθίσει σε περισσότερες καινοτομίες από αυτές που εσείς ε, μας λέτε. Τώρα, πιο σοβαρά. Σας ακούω και ακούω τα ίδια. Δηλαδή, ότι αν ο στόχος μας είναι περισσότερο ΕΠ, με μια πράσινη συνιστόσα, βλέπουμε ότι οδηγεί σε δύο πράγματα. Πρώτον, περισσότερες διαφορές μεταξύ του κόσμου και περισσότερη κατανάλωση των ε, πηγών ενέργειας που έχουμε στον πλανήτη μας. Οπότε η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Εσείς τι θα αλλάζατε σαν οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, γιατί όταν σας ακούω είναι σαν να λέτε ότι ε, θέλετε λιγάκι να το προσαρμόσετε, αλλά όχι να το αλλάξετε. Θα αλλάζατε κάτι αν αυτό εξαρτιόταν από εσά. Ευχαριστώ. Μιλάτε με κάποιον που πρώτος έβαλε το θέμα αυτό, που πάει βέβαια μπρος πίσω. Θέλω να πω με αυτό ότι εδώ βέβαια υπογραμμίζεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και εγώ νιώθω απόλυτα δεσμευμένο σε αυτό που λέτε εσείς την πράσινη συνιστόσα και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για μία ολόκληρη διάσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πρασίνισμα των πολιτικών μας. Η φορολογία που συζητάμε στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ φιλόδοξοι όσον αφορά την πράσινη αυτή διάσταση. Θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα στο 20% και να αυξήσουμε κατά 20% τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και τις ανανεώσιμες. Πρόκειται λοιπόν για συνδυασμό νομοθεσίας και φορολογίας από τη μια και από την άλλη μεριά καινοτομία και τεχνολογίας. Είναι πράγματα που πάνε μαζί. Οι πολιτικοί πρέπει να διασφαλίσουν και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι υπάρχει η δυναμική που χρειάζεται για να επιτευχθεί το νομοθετικό έργο και να προχωρήσει η τεχνολογία ώστε να έχουμε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο της κοινωνίας μας. Γίνονται πράγματα, αλλά σίγουρα μένουν και πολλά ακόμα να γίνουν. Μην αμφισβητείτε όμως τη δικιά μου τη δέσμευση υπέρ αυτής της πράσινης διάστασης. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο συγκεκριμένος όσον αφορά την αντικατάσταση του ΕΠΟ ω δείκτη η, χρήση ενός άλλου πιο πλούσιου δίκτυ για να δούμε ποια είναι πραγματικά η αξία της ανάπτυξης. Εσείς πού βρισκόσαστε ακριβώς στα πλαίσια όλης αυτής της συζήτησης. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη. Θέλετε να απαντήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, πού βρίσκομαι. Όχι στη μέση, αλλά και στις δυο πλευρές. Δηλαδή, πιστεύω ότι χρειάζεται ένα δείκτης μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπω είναι το ΕΠ, και που να είναι ένας παγκόσμιος δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας, και λειτουργεί αρκετά καλά για το σκοπό αυτό. Βέβαια, πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται βάσει του στατιστικού συστήματος. Συγχρόνως, όμως λέω ότι για το λόγο για τον οποίο το χρησιμοποιούμε, λειτουργεί καλά. Συγχρόνως, πέρα από το ΕΠ και στις γραπτές μου απαντήσεις θα το δείτε ότι σκοπεύω να υποβάλω πρόταση, από κοινού με τους συνεδέρφους βέβαια, για ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που να μετράει στατιστικά με άλλους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης. Όχι μόνο δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη, αλλά να μπορούμε να μετρήσουμε και άλλους παράγοντες ανάπτυξης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να μετρήσει την ευτυχία του ατόμου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείχτης για την ευτυχία του ατόμου. Κύριε Φόρτ τώρα. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίθασατε σε αυτή την επιστροπή. Αναφερθήκατε στο δυσβάχστατο δημόσιο χρέος και τη, δυνα... και τη σημασία να επενδύσουμε στην καινοτομία για την ανάπτυξη. Σύμφωνο με αυτά. Και μετά περιγράψατε νέα εργαλεία του δημόσιου τομέα για τις επενδύσεις. Και αυτή η ισορροπία μου θυμίζει μία Βρετανίδα πολιτικών πριν από μερικές δεκαετίες που έλεγε δεν μπορείτε να ξοδεύετε χρήματα που δεν έχετε. Μήπως αυτό θα ξανασυζητήσουμε. Ελπίζω όχι. Όταν ήρθε όμως στην Επιτροπή αυτό ο κύριος Μόντι και περιέγραψε τις επενδύσεις και την έρευνα, είπε ότι οι αποδόσεις είναι το βασικό κίνητρο και η Ευρώπη έχει μόνο 50% της έρευνας που χρηματοδοτείται από αυτές τις πηγές. Στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία είναι πολύ υψηλότερα. Και είπε ο κύριος Μόντι ότι δεν πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους γιατί αυτό θα μειώσει τις επενδύσεις στην έρευνα και ότι μέσω πρόθεσμα θα πρέπει να επιδιώκουμε μείωση των φόρων. Εσείς τι πιστεύετε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αναμένω την νέα έκθεση του Μάριο Μόντι για την περάτωση της ενιαίας αγοράς που θα παρουσιάσει τον Απρίλιο. Είχα κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις μαζί του και αναμένω την τελική του έκθεση. Βεβαίως, μια και αναφερθήκατε στον Μάριο Μόντι και εσείς και αυτός έχετε δίκιο ότι ο ιδιωτικός τομέας σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες για μεγάλο τμήμα είναι ο υπεύθυνο για την επενδύσει στην έρευνα και στην καινοτομία. Και ένα από τα διδάγματα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα δημόσια μας οικονομικά δεν θα επιδεινωθούν έτσι ώστε να διώξει τις ιδιωτικές επενδύσεις, πράγμα το οποίο θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητά μας να επενδύσουμε σε έρευνα και κοινοτομία. Γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτά που είπα στην αρχή και συγγνώμη αν φαινομαι επίμονος. Πιστεύω ότι βιώσιμα δημόσια οικονομικά και επενδύσεις στην απασχόληση και στην βιώσιμη οικονομική είναι μαζί και αυτά είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε μετά και τις επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία. Follow Την πληρωματική ερώτηση. Μπορείτε να μου απαντήσετε για το τι πιστεύετε για την άποψη του κυρίου Μόντι ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να έχουμε ακόμα επενδύσεις από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί και οι φόροι που τους επιβάλλουμε. Η απάντησή μου είναι απλή. Ναι, και εγώ ο ίδιος ασχολήθηκα με δύο φορολογικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μου όταν αντιμετωπίσαμε τη χειρότερη μας οικονομική κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικά φορολογικά συστήματα που να είναι και δίκαια και να υποστηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Ρεν, ομολογώ ότι είχα ετοιμάσει άλλη ερώτηση να σας κάνω. επειδή όμως είναι πρόσφατη η επίσκεψη κλιμακίου της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα, αναφερθήκατε κι εσείς, οφείλω να σας πω ότι αυτή η επίσκεψη συγκέντρωσε δικαιολογημένα την οργή της κοινή γνώμης. Γιατί? Διότι οι απεσταλμένοι σας, κατά την εξευθελιστική διαδικασία στην οποία υπέβαλαν τους υπουργούς, μίλησαν για περικοπή των μισθών και ισχυρίστηκαν ότι μία σύνταξη των 720 ευρώ είναι αρκετή και πρέπει να περικοπεί. Καμία ερώτηση από τους αποσταλμένους σας, βάσει των στοιχείων που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και αλλού, Επίσης πρότειναν μείωση των συντάξεων τη στιγμή που υπάρχει εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή από τις επιχειρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και ε, ε, απώλεια εισφορών από το θέμα της ανασφάλισης εργασίας. Σας ερωτώ λοιπόν, το οικονομικό πρόβλημα είναι θέμα δαπανών, δεν είναι θέμα εσόδων. Τι γνωρίζετε αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνετε στο ζήτημα αυτό και ιδιαίτερα στο ζήτημα της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής. Uh, Κοιτάξτε, η φοροδιαφυγή είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπουδήποτε υπάρχει και ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραθυράκια γιατί αυτά αποδυναμώνουν τη φορολογική βάση των δημόσιων και των κοινωνικών υπηρεσιών μας. Αυτών όλων λεχθέντων πρέπει να πω ότι το θέμα μου σε αυτά τα φορολογικά είναι κατ' ουσίαν αρμοδιότητα των κρατών μελών τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή. Ως εκ τούτου, σε αυτή την περίπτωση, οι ελληνικές αρχές θα έλεγα ότι είναι εκείνες που φέρουν την ευθύνη για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τόσο τη φοροδιαφυγή, όσο και το να διασφαλίσουν την λειτουργία, την αποτελεσματική λειτουργία των λογιστικών τους στο μέλλον. Συμπληρωματική ερώτηση. Με ποια ισχύ με ποια εντολή, δεν ξέρω αν ήταν από τον κύριο Αλμούνια ή από εσά, κατά τα άλλα οι απεσταλμένοι σας έκαναν υποδείξεις στον τομέα των συντάξεων ή και στον τομέα των μισθών. Σας έχουν ενημερώσει. Γιατί δεν περιμένετε την ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει το πρόγραμμα σταθερότητα παρά δίδετε στη δημοσιότητα τι ακριβώ ζητούν και μάλιστα απεσταλμένοι σα έναντι υπουργών. right that... Uh, Έχετε δίκιο ως προς το ότι πράγματι πρέπει να περιμένουμε την ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει το πρόγραμμα σταθερότητας. Πρέπει να περιμένουμε ένα ε, περιεκτικό και πιστικό πακέτο το οποίο θα περιλαμβάνει χειροπιαστά μέτρα τα οποία θα ανοίξουν το δρόμο για να περιοριστεί το υπερβολικό έλλειμμα μέχρι το όριο που προβλέπεται στα κριτήρια σταθερότητας. Βεβαίως, εν ευθέτω χρόνο. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές και μόλις κατατεθεί το πρόγραμμα σταθερότητας κάποια στιγμή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις ε, στην Επιτροπή είτε στην ΝΙΝ είτε στη Μελλοντική Επιτροπή. Προχωράμε τώρα στην, ε, στον επόμενο μιλητή από τους, στην ομιλήτρια μάλλον στην κυρία Αντρέσεν από τους Ελεύθερους Δημοκράτες. Από ό,τι φαίνεται η ένταξη, η συμμετοχή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν υπόφοροι για ορισμένα κράτη-μέλη. Όταν εισήχθη το ευρώ αυξήθηκε αυξήθηκαν κατά πολύ οι τιμές ε, στην Ευρωζώνη και στην Εστονία το 75% φοβούνται ότι αν ε, υιοθετήσουν το ευρώ θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές. Κάτι τέτοιο προβλέπεται για του χρόνου. Συμφωνείτε ότι το να υιοθετήσει κανείς το ευρώ οδηγεί αυτόματα σε ανατιμήσεις. Και τι προτείνετε. Ε, προτείνετε να υιοθετήσουν και άλλες χώρες το ευρώ. Και επόμενη ερώτηση οι χώρες που πρέπει να υποτιμήσουν το νόμισμά τους για να αντιμετωπίσουν την οικονομική και νομισματική κρίση και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Τι πρέπει να κάνουν? Ε, θα απαντήσω στην ερώτηση στην πρώτη. Εκεί θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μου. Όσον αφορά τις ε, ανατιμήσεις, αυξήσεις τιμών. Κοιτάξτε, η συμμετοχή στην Ευρωζώνη δεν πρέπει να οδηγεί σε αυξήσεις τιμών. Βεβαίως, τούτο είναι συνάρτηση της οικονομικής πολιτικής της κάθε χώρας και της ε, ικανότητάς της να ανταπεξέλθει στο χαμηλό πληθωρισμό και αυτό είναι ένα από τα κριτήρια για να μπει μια χώρα στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχουν ε, σημαντικές ενδείξεις ε, για ανατιμήσεις έστω και αν υπάρχουν κάποιες ε, μικρές αυξήσεις τιμών, όταν γίνεται το περίφημο στρογγύλεμα της τιμής, αλλά αν τελικά η οικονομική πολιτική είναι ε, σωστή και υπάρχει συγκράτηση του πληθωρισμού, δεν θα πρέπει το ευρώ να οδηγεί σε ανατιμήσεις. Ρωτήσετε κατά πόσον είμαι υπέρ ή κατά της διεύρυνσης της ε, ευρωζώνης. Εγώ είμαι υπέρ με βάση τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όταν μια χώρα καλύπτει, πληρεί τα κριτήρια για την Ευρωζώνη, επόμενος υποψήφιος είναι η Εστονία, θα πρέπει να της δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Η Εστονία κοντά είναι στην Ευρωζώνη, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σέβεται τους κανόνες, σέβεται τις συνθήκες και στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε την άνοιξη στην έκθεση περιστονίας για το κατά πόσον καλείται κριτήρια σύγκλησης. Κύριε Ρεν, η Σλοβακία έκλεισε ένα χρόνο στην ε, Ευρωζώνη και βίωσε μεγάλες ανατιμήσεις, μέχρι και 25%. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά άλλο ένα, της, ε, κατά 1% περισσότερο από ότι της ε, Τσεχίας. Πώς μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε, πώς λέτε ότι η εισαγωγή του ευρώ δεν επηρεάζει τις τιμές. Ε, κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία που μα αναφέρετε μπορούν να εξηγηθούν με διάφορους τρόπους. Πάντω, η Σλοβακία, εγώ έχω πολλούς φίλους στη Σλοβακία και σας λέω ότι η πλειοψηφία αυτών με βάση του γνωστού μου πάντα, είναι δική μου η σφιγμομέτρηση, αυτοί είναι ικανοποιημένοι που μπήκαν στην Ευρωζώνη. Το ευρώ τους ε, προστάτευσε από τη θύελα της ε, οικονομικής κρίσης Τη Σλοβακία την ξέρω πολύ καλά ως χώρα. Θυμάμαι πολύ καλά ε, την ε, ύφεση στις αρχές της δεκαετίας των 90. Τότε η Φινλανδία δεν είχε το ευρώ και εμείς ε, υποφέραμε πάρα πολύ από την ενεργεια, Τεράστιο το ανθρώπινο κόστος. Και τώρα έχουμε το ευρώ, το οποίο προστατεύει και μεγαλύτερα και μικρότερα κράτη-μέλη μεσούσεις της θέλης της οικονομικής κρίσης. Επιστρέφουμε στο ΕΛΚΟ. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο. Oh, uh, Κύριε Ρεν, βλέπουμε ότι έχετε καλή θέληση, καλές προθέσεις, αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν έχετε και τις απαραίτητες αρμοδιότητες ε, ε, λόγω ε, του ότι υπάρχει τέτοιο κενό και έχουν γίνει και σχετικές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια. Όπως και σε όλους τους άλλους τομείς ε, πρέπει να επιδείξετε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ηγετικά καθήκοντα. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, τους στόχους που αναφέρετε δεν πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να τους επιτύχουμε καλύτερα εφόσον η Κομισιόν υποβάλλει ένα συγκεκριμένο κατάλογο για μέχρι το 2020 και να πει σε κάθε κράτος μέλος το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ποιοι είναι οι αριθμοί, πώς ελέγχονται οι αριθμοί και ερωτώ, είσαστε πρόθυμος να συστήσετε μια επιτροπή διαμεσολαβητική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική εξόδου. Γιατί το έλλειμμα είναι εκείνο που μπορείτε να επέμβετε στο έλλειμμα. Μπορείτε και να επιβάλλετε κυρώσεις και να επιβραβεύσετε. Τι ακριβώς σκέφτεστε γύρω από όλα αυτά. Κατά τη δική μου άποψη, το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη μοιάζει με μία συμφωνική ορχήστρα. Δηλαδή, όλοι οι μουσικοί πρέπει ε, να συντονίζονται για να επιτύχουν τον κοινό στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Να συνεργαζόμαστε λοιπόν και κατά την άποψή μου ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 της πολιτικής αυτής όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ε, ανεργία, ο καλύτερος τρόπος είναι όλοι μαζί να ορίσουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους που να αφορούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά Μπορούμε βέβαια να δούμε ε, πώς κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιδιώξει αυτούς τους στόχους και να βάλει και τους δικούς του. Και 27 πρέπει να έχουν τον ίδιο ευρωπαϊκό στόχο. Και αυτά θα τα επιτύχουμε μέσα από την επιτήρηση αλλά και μέσα από την ανέβρεση νέων εργαλείων για να χρηματοδοτήσουμε όλους αυτούς τους ε, τόσο σημαντικούς στόχους. Κατά την άποψή μου, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον. Δηλαδή, συνδυασμός ε, συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, ε, ολοκλήρους κοινή αγοράς, κοινοτικέ δηλαδή αποφάσεις και καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία έτσι ώστε να βρούμε τους πόρους τους πόρους που θα είναι απαραίτητοι για να υπάρξουν επενδύσεις και να εφαρμοστεί η στρατηγική εξόδου. Συμπληρωματική ερώτηση από αυτού. Ως εκ τούτου δηλαδή θα, ήταν, θα είχε νόημα να είχαμε και έναν κοινό, κοινοτικό ισολογισμό. Γιατί σε πολλέ περιπτώσεις δεν ξέρουμε κατά πόσον ευσταθούν τα στοιχεία που μα δίνουν τα κράτη-μέλη. Ε, είναι διαφορετικές και εξολογήσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεωρείτε κι εσείς ε, ότι για να υπάρχει αυτή η νέα συνεργασία είναι να, υπάρξει και νέ, να υπάρξουν νέοι ισολογισμοί που θα κατατεθούν έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συντονισμός. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτησή σας, η οποία υπάρχει στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ τα θυμάμαι αυτά ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ήδη από τα μέσα της δεκαετίας των 90. Ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά ενδελεχώς και θα γίνει κάτι τέτοιο ε, στο πλαίσιο της ε, ενδιάμεσης δημοσιονομικής αναθεώρησης που θα ανοίξει το δρόμο για τη δημοσιονομική προοπτική για το, μέχρι το 2014. Ενδιάμεση αναθεώρηση συν ε, στόχοι για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Κατά την άποψή μου, οι στόχοι της πολιτικής 2020, καινοτομία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες, αυτά πρέπει να προβληθούν στο πλαίσιο της ε, δημοσιονομικής αναθεώρησης. Και κατά την άποψή μου, ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξυπηρετεί καλύτερα τις επενδύσεις για να υπάρχει περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο πράσινη και περισσότερο ευφύης οικονομία. Η επόμενη ερώτηση, κύριος Κάρεν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, πέρασαν 8 χρόνια από τότε που έχουμε το ευρώ και 5 χρόνια από τη πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 όμως από τις 27 χώρες μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης. Και από αυτές 8 είναι από τις καινούργιες χώρες μέλη. Ρωτάω λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς την παρετέρω διαδικασία όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωζώνης και ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπετε εσείς για αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Εποφελούμε και εγώ από την ευκαιρία για να μιλήσω κι εγώ τη μητρική μου γλώσσα. Δεν θέλω να το ξεχνάω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θέτεται. Και όπως είπατε, 11 από τις 27 χώρες μέλη δεν είναι ακόμα μέσα στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη έχει δείξει τα τελευταία δέκα χρόνια τι μπορεί να κάνει, τη δύναμή της. Αν μη τι άλλο, τώρα τελευταία με την οικονομική κρίση και την ύφεση που είχαμε. Το ευρώ μας προστάτευσε από τη θύελα όχι μόνο τις μικρές χώρες μέλη, αλλά και τις πιο μεγάλες. Και ακριβώς γι' αυτό καταλαβαίνω πολύ καλά που πολλές από τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν και να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Βάσει της συνθήκης, αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε καλά αποτελέσματα, μακροοικονομική σταθερότητα και υπάρχουν πέντε συγκεκριμένα κριτήρια για να αξιολογηθεί αυτή. Επίσης, εκτιμάμε κατά πόσο μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι ακόμα μέλος στην Ευρωζώνη μπορεί με επιτυχία να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Η υποψήφια χώρα που προβλέπεται πρώτη να μπει στην Ευρωζώνη είναι η Εστονία. Τα αποτελέσματα εκεί, οικονομικά, είναι αρκετά καλά και όσον αφορά το χρέος. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω όμως να τονίσω ότι όσον αφορά την Εσθονία ε, θα συμμορφωνόμαστε πλήρως τους ε, κανόνες και η χώρα θα συμμορφώνεται σε όλα τα κριτήρια για να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Εντάξει, και εγώ θα κάνω αυτό το γλωσσικό πινκ-πονγκ ε, αγγλικά θα θέσω τη συμπληρωματική μου ερώτηση. Τα κριτήρια του Μάστριχτ. Όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωζώνης. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι περισσότερες από τις χώρες που είναι τώρα στην Ευρωζώνη παραβιάζουν ή ένα ή και πολλά κριτήρια από τα κριτήρια σταθερότητας. Οπότε, ποια είναι η γνώμη σας. Ξέρουμε ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε αποτελεί συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης. Είναι πολύ βασικό όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να επανέλθουν σε υγιή δημοσιονομικά. Το είπα και το ξαναείπα σήμερα το βράδυ αυτό, ότι αυτό θα είναι ένα από τα κύρια καθήκοντά μου εφόσον τελικά οριστώ Επίτροπος Αρμόδιος για τα Οικονομικά Ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πέντε κριτήρια ήταν πάντα δείκτες για να ξέρουμε κατά πόσο μία χώρα μπορεί να έχει σταθερά δημοσιονομικά, αλλά και κατά πόσο έχει την πολιτική βούληση ώστε να υπάρξει αυτή η σταθερότητα και να τηρηθεί. Είναι και αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Εσέα τώρα. Η κυρία Εσέα. Ευχαριστώ κύριε Ρεν. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ τη μητρική μας γλώσσα, τα φιλανδικά, οπότε και εσείς, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φιλανδική γλώσσα για να μου απαντήσετε. Είναι γνωστό γενικά ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να φέρουν σε πέρα στις υποχρεώσεις τους, κάτι το οποίο μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες και να πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μέτρα για να μας βοηθήσουν, μάλλον για να βοηθήσουν τα κράτη αυτά μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους αυτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για οικονομικές αναλύσεις και οικονομικά στοιχεία που δίνουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να παίρνει αξιόπιστα στοιχεία, στατιστικά δεδομένα από τις διάφορες χώρες. Μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σωστά στοιχεία, αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα είναι αυτό που αποτελεί και τη βάση της σωστής οικονομικής ανάλυσης και ένα των σωστών ε, αποφάσεων που θα πάρουμε. Άρα δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι ένα θεσμικό πρόβλημα. Και υπάρχουν πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό η Ελλάδα και το δημόσιο της έλλειμμα σε τι βαθμό έχει μεγαλώσει, πόσο και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο μακροπρόθεσμα να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Βραχυπρόθεσμα εντάξει, ξέρουμε ότι σαφώς και υπάρχει ανάγκη για πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που θα έχουν άμεσα κάποιον αντίκτυπο έτσι ώστε να βγει από το έλλειμμα αυτό η χώρα. Ξέρουμε ότι είναι αναγκαία μια διόρθωση. η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε να παίρνει μέτρα και η Επιτροπή και η Eurostat στηρίζουν την Ελλάδα στα μέτρα αυτά που παίρνει προκειμένου τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας έρχονται από εκεί να είναι σωστά και αξιόπιστα. Πριν από τέσσερα χρόνια στην παρουσίαση της Επιτροπής ζητήθηκε έλεγχος. Το Συμβούλιο όμως δεν συμφώνησε με την απόφαση του 2005 γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να το ξαναδούμε. Και θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει τέτοιες εξουσίες ελέγχου προκειμένου να ε, διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που μας έρχονται από τα κράτη-μέλη είναι αξιόπιστα. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Ναι, με σαφήνεια είπατε ότι θέλετε να επικεντρωθείτε στη Eurostat και στα στατιστικά δεδομένα που μας έρχονται από τα κράτη-μέλη, προκειμένου αυτά να είναι σωστά και αξιόπιστα. Προβλέπετε τίποτα κυρώσεις, σκέφτεστε τίποτα κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε χώρες μέλη, εφόσον αυτές επανειλημμένα δίνουν λάθος ή μη αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Ο κύριος Ρεν. Υπάρχει η κοινοτική υπαρχει η κοινοτικη νομοθεσια που προβλέπει ποινικέ κυρώσεις εφόσον ε, κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχουν δυσλειτουργίες. Αυτό όμω που μα ενδιαφέρει μα πάνω απ' όλα είναι τα διορθωτικά μέτρα. Μέτρα δηλαδή τα οποία βοηθούν να διορθωθεί η κατάσταση σύντομα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την ελληνική κυβέρνηση, με τις ελληνικές αρχές. Εμείς στηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειέ τη να διασφαλίσει αξιόπιστα και σωστά στατιστικά στοιχεία που να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κοινοτικές απαιτήσεις στους... Yes, thank uh, Κύριο Σικλούνα. Κύριε Ρεν, ήδη οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ότι δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στους δύσκολους καιρούς. Και απαντήσατε ότι θα εξετάσετε περαιτέρω τον συντονισμό και την εποπτεία των δημοσίων οικονομικών πολιτικών. Αλλά επανέρχομαι στο θέμα των στατιστικών. Γιατί πιστεύω ότι η αξιοπιστία διακύβευεται όταν πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν μια πραγματική ανεξάρτητη αρχή για στατιστικά στοιχεία. Δεν έχουν χρηστή διακυβέρνηση για τα στατιστικά στοιχεία. Και αναφερθήκατε σε δύο αποτυχίες σε μια συγκεκριμένη χώρα, Λέμε σίγουρα ότι κι άλλες θα ανακαλυφθούν. Μήπως πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποιο είδους απαιτήσει εποπτείας. Παραδείγματος χάρη. Πολλές κυβερνήσεις εκδίδουν υπερβολικά αισιόδοξε προβλέψεις, πράγμα το οποίο μετά έχει αλυσιδωτές επιδράσεις στα δημόσια τους οικονομικά. Μήπως πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και για την μεσοπρόθεσμη διακυβέρνηση των οικονομικών από τα κράτη-μέλη. Απάντηση. Ζήτησα μάλιστα από τους συνεργάτες μου να μελετήσουν την περίπτωση της Ελλάδος σε ό,τι αφορά το στατιστικό της σύστημα και τη λειτουργία του. Και επίσης ζήτησα πληροφορίες για τα άλλα κράτη-μέλη. Και οι πληροφορίες που έλαβα λένε ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική περίπτωση και τα προβλήματα είναι πράγματι πολύ σοβαρά όπως αναφέρονται και στην έκθεση της Κομισιόν που υιοθετήσαμε την Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η ε, σωστή λειτουργία του στατιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Για την περίπτωση της εισόδου στο ευρώ, της προσχώρησης στο ευρώ της Σλοβακίας. Θα θυμάστε ίσως, αλλά σας το θυμίζω, ότι η Σλοβακία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό έλεγχο από την Ευρωστάτ για το δημόσιο της έλλειμμα. Η Ευρωστάτ με αποστολές αξιολόγησε πράγματα όπως το πώς κάποιες επενδύσεις σε υποδομές ή κάποιες δαπάνες νοσοκομιακές ταξινομούνται στους δημόσιους λογαριασμούς της Σλοβακίας. Και αυτό το παράδειγμα μας ενεθάρρυνε. Γιατί έμαθα πολλά πράγματα από διάφορες πηγές. Τέτοιου είδους αυστηρότητα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να εξασφαλίσουμε ότι τα στατιστικά μας στοιχεία θα είναι σωστά σε εθνικό επίπεδο και η Ευρωστάτ να κάνει και αυτή τη δουλειά της για να εξασφαλίσει ότι το όλο σύστημα είναι υπόλογο και δουλεύει αξιόπιστα. Συμπληρωματικό ερώτημα. Πώς θα επιτύχουμε ισορροπία, γιατί η, η Κομισιόν είναι πολύ σοβαρή με τέτοιου είδους ελλείψεις, αλλά δεν θέλουμε η ίδια η Κομισιόν να τα κάνει όλα αυτά από μόνη της. Και αυτό και για τους φορολογικές κανόνους. Γιατί υπάρχουν πολλές καλές χώρες που λειτουργούν σωστά, που έχουν καλούς φορολογικούς κανόνες και μπορούν να καθορίσουν ένα μέσο πρόθεσμο φορολογικό πλαίσιο από μόνες τους. Απάντηση. Κατά την άποψή μου, μπορούμε να θίξουμε το θέμα αυτό στα πλαίσια της, ε, του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και της εποπτείας. Αρχικά, συζητήσαμε την δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των δημοσίων οικονομικών της Ευρωζώνης και μάλιστα των άλλων κρατών μελών εκτός Ευρωζώνης στα πλαίσια των προγραμμάτων σύγκλησης και σταθερότητας. Ένα από τα διδάγματα αυτής της κρίσης είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε μέσο πρόθεσμα και να λάβουμε δράση βράχη πρόθεσμα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δημόσια οικονομικά είναι βιώσιμα. Κύριος Πέντα. Äh, Στην ε, συνάντηση με τον ε, κύριο Μπαρόζο, ακούσαμε τον κύριο Μπαρόζο να υπόσχεται ότι θα λάβει περαιτέρω μέτρα όσον αφορά στην οδηγία πλαίσιο ε, για υπηρεσίες καθολικού συμφέροντος. Ε, μήπως έχετε λοιπόν μια ε, σαφέστερη εικόνα ή ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει αυτή η εργασία. Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την επόμενη Κομισιόν και χαίρομαι που ο πρόεδρος κ. Μπαρόζο υπογράμμισε τόσο στεναρά αυτά τα θέματα όπως έγινε και κατά την προετοιμασία των ακροάσεων που έλαβε χώρα την Πέμπτη. Εγώ προσωπικά ε, θέλω να καταθέσω πιστικές προτάσεις για να υπάρχει ένα ποιοτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Βεβαίως ε, δεν είναι άμεση δική μου αρμοδιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα αποφασιστεί από το σύνολο των επιτρόπων αλλά κατά την άποψή μου η πρόταση αυτή πρέπει να κατοτεθεί κατά τη διάρκεια αυτού του έτους τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο. Και συμπληρωματική ερώτηση. Νομίζω δεν υπάρχει επιλογή. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περικόψουμε τις δημόσιες δαπάνες και για να μπορούμε να παραμείνουμε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που το 2008 εμείς στην Εστονία κατορθώσαμε να παραμείνουμε στο 2,75% όσον αφορά το έλλειμμα και 3,1%. Αυτό ανήλθε στο 3,1 το 2009. Βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θέλω να ξέρω το δικό σας το όραμα όσον αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ποια θα πρέπει να είναι η σωστή στρατηγική της Βαλτικής για να υπάρχουν και οι καλές συνεργασίες. Βεβαίως και τα κράτη-μέλη φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη, αλλά η περικοπή των δημόσιων δαπανών μήπως είναι κάτι που μπορεί να ακολουθηθεί και στη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, όσον αφορά την Εστονία, το φυσικό πλαίσιο ε, για, την, για το συντονισμό είναι η Ευρωζώνη, όταν η Εστονία μπει στην Ευρωζώνη. Με βάση βέβαια τους κανόνες όπως να ακολουθεί και εφόσον πληρεί τα κριτήρια. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας ε, για τις χώρες της Βαλτικής, ε, παραδείγματο χάρη ε, σε περιβαλλοντικά θέμα, θέματα, αλλά και σε θέματα ναυτιλιακά, θέματα επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ένα καλό παράδειγμα που συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία είναι τα κονδύλια που εδόθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει συνεργασία στις χώρες της Βαλτικής. Η Εστονία είναι χώρα κλειδί και κύριος αποδέκτης αυτών των επενδυτικών κονδυλίων. Περνάμε στους φιλελεύθερους, ο κύριος Τρεμόσα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ρεν, επικεφαλής ε, του Ευρωπαϊκού ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα εφόσον η Ελλάδα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήσει βοήθεια. Πιστεύετε εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει έναν μηχανισμό προκειμένου να βοηθάει χώρες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και πιστεύετε ότι διορθωτικά μέτρα θα έπρεπε να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη τα οποία δεν ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ. Απάντηση. Μιλάμε για διαχείριση κρίσεων στην περίπτωση προβλημάτων με τα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι ένα άλλο και άλλη είναι η βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια χώρα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τη γνώμη μου, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει εξορισμού να διασφαλίζει ότι οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης έχουν υγιή δημόσια οικονομικά τηρούν τους κανόνες του συμφώνου και κατά γράμμα και κατά το πνεύμα. Άρα δεν χρειάζεται τέτοιο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων. Δεν χρειάζεται τέτοιο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων κανονικά. Τώρα βέβαια πρέπει να επικεντρωθούμε στην σωστή εφαρμογή του συμφώνου και πώς θα φροντίζουμε να γίνεται αυτή η σωστή εφαρμογή του συμφώνου, πώς θα επιβάλλουμε τη σωστή εφαρμογή του συμφώνου. Έχουμε την περίπτωση της Ελλάδας και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με την ελληνική κυβέρνηση και περιμένουμε το ε, συνολικό τελικό ε, σχέδιο της Ελλάδας, την πρόταση της Ελλάδας, το πακέτο το οικονομικό που θα προτείνει η Ελλάδα για να βγει από, από το πρόβλημα αυτό. Τώρα από την άλλη, αν δεχτούμε κάποιες αρχές. Ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός εξάντε. Επιμονή μου βάσεως. Για τέτοιες περιπτώσεις, για να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις, είναι κάτι που μπορούμε να δούμε. Συμπληρωματική ρώτησε Ο κύριο Τρισέ πριν από ένα μήνα περίπου ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να εφαρμόσει ειδικέ πολιτικέ για ειδικέ ε, χώρε που αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στην Ευρωζώνη. Είπε ότι η Ελλάδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Εσεί πιστεύετε ότι τα ευρωομόλογα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τι χώρε τη Ευρωζώνη να αντιμετωπίσουν την κρίση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τρισέ ότι υπάρχει ένα ευρώ, άρα ενιαία νομισματική πολιτική. Ο κύριος στόχος τώρα, ο πρώτος και κύριος στόχος μας είναι η σταθερότητα, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης να εφαρμόζεται πραγματικά με τρόπο τέτοιο που να αποφεύγει περιπτώσεις μη υγιών δημοσίων οικονομικών. Για να μην χρειάζονται μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσης. Απάντησα πριν την ερώτησή σας για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Νομισματικού Ταμείου και είπα ότι όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε με ανοιχτό πνεύμα, αλλά όχι να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσης. Γιατί τίθεται και ηθικό ζήτημα εκεί. Ευχαριστώ από τους Πρασίνους. Κύριε Ρεν, αναφερθήκατε στο ανοιχτό σας και καινοτόμο πνεύμα. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για φορολογική συνεργασία, γιατί εξ αρχής μιλάτε για την αναγκαιότητα υγιών δημοσίων οικονομικών, αλλά δεν μιλάτε για τα μέσα να το πετύχετε. Υπάρχουν δύο μεγάλα μέτρα να συνεργαστούμε για τις δαπάνες ή να καταπολεμήσουμε από κοινού τις ε, φοροδιαφυγές. Η Κομισιόν λέει ότι χάνονται 200 δις σε ε, φορολογικούς παραδείσους. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μειώνεται η συνεισφορά των φορολογουμένων για αυτές τις δαπάνες εξαιτία της φοροδιαφυγής. Όμως εσείς ως Επίτροπος που είστε υπεύθυνο για την μακροοικονομική σταθερότητα και την υπεύθυνο για καταπολέμηση των ελλημάτων, τι θα προτείνετε στην θητεία σας. Ευχαριστώ. Θα συνεργαστώ βεβαίως με τον συνάδελφό μου, τον προτινόμενο Επίτροπο κύριο Σεμέτα για θέματα φορολογικού χαρακτήρα και σωστά είπατε ότι με ενδιαφέρει το θέμα και εσάς επίσης σας ενδιαφέρει γιατί ως μέλη αυτής της Επιτροπής και ως Ευρωπαίους φορολογούμενους θα πρέπει όλοι να προσπαθούμε να κλείσουμε τα παραθυράκια και να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Κατά την άποψή μου λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας οι οποίες κατά κάποιο βαθμό έχουν προοδεύσει τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια στα πλαίσια της ομάδας των 20 για να έχουμε υγιείς διεθνείς κανόνες κατά των φορολογικών παραδείσων. Το βασικό, κατά την άποψή μου, είναι ένα υγιές και σωστό διεθνές φορολογικό καθεστώς δεν συμπεριλαμβάνει φορολογικούς παραδείσους. Είδαμε τα τελευταία χρόνια μεγάλες κινήσεις κεφαλαίων και δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους τάσεις είναι καλές για την βιώσιμη απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών. Η Κομισιόν εργάζεται και θα εργαστεί κατά της επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού. Η μείωση της φορολόγηση είναι εθνική αρμοδιότητα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε για χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμό των διεθνών κανόνων στον τομέα αυτό. Και για να τελειώσω, τον Οκτώβριο πέρυσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσει μία πιθανή συνεισφορά των καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τελών για, τις, ε, για τα επενδυτικά κεφάλαια. Θα το διερευνήσουμε αυτό και κατά τη διάρκεια της Άνοιξης και θα συζητήσουμε και θέματα που σχετίζονται με διεθνή φορολογικά καθεστώτα. Συμπληρωματικό ερώτημα για τις καινοτόμες λύσεις που απαιτούνται. Τι πιστεύετε εσείς για την πρόταση που είχε υποβάλει η Κίνα στη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου για μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος και την ιδέα να πάμε προς ένα πιο συστηματικό να μεταβούμε προς ένα πακέτο νομισμάτων ε, για να φύγουμε από το δολάριο. Απάντηση. Το θεωρώ ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο το ότι η Κίνα είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε πολυμερή συντονισμό για έλεγχο των νομισματικών πολιτικών και των ισοτιμιών. Το είδαμε αυτό και στα πλαίσια της ε, ε, κρίση στο τέλος του 2008 όταν όλες οι μεγάλες τράπεζες, η έκτη, η, τράπεζα της Κίνας από κοινού αντιμετώπισαν τα επιτόκια. Κατά την άποψή μας η, το, η ισοτιμία του ευρώ και σε σχέση με το δολάριο και με του Γιάν είναι πιθανός κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους Κινέζους για το θέμα και διμερός και πολυμερός. Ε, thank you. Um, ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντ ξανά. Ζητώ συγγνώμη κάποιοι συνάδελφοι ασθενούν. Μερικές φορές η Βρετανία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Ξανά θα μιλήσω για μεγάλα ελλείμματα. πολλοί αναφερθήκαμε στην Ελλάδα, αλλά η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Λετωνία, πολλές άλλες χώρες, η Ιρλανδία και αυτές έχουν μεγάλα ελλείμματα. Θα ήθελα κυρίως να καταλάβω τη δική σας άποψη για το βρετανικό έλλειμμα και την εμπιστοσύνη σας για το τι μέτρα θα λάβει η Βρετανική κυβέρνηση και τι πιστεύετε για όλα αυτά τα χρέη που είναι εκτός του ισολογισμού. Ξέρω ότι και άλλες χώρες πέραν της Βρετανίας έχουν τέτοιου είδους χρέη. Thank you. Thank you, Σας ευχαριστώ, κυρία Φόρντ. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω την πρόθεση να συμμετάσχω στην εσωτερική πολιτική συζήτηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή ούτε σε οποιοδήποτε συζήτηση άλλου κράτους μέλους. Κάνω τη δουλειά μου απλώς. Για να έχουμε υγιή δημόσια οικονομικά στην Ευρώπη. Υπάρχει μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αναμένουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να μειώσει το έλλειμμά του για να σεβαστεί και τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα όπως ξέρετε πολύ καλά και για να είναι επιτυχές αυτό το χρονοδιάγραμμα πρέπει να υπάρξει ε, κάποια ετήσια μείωση του δημοσίου ελλείμματος. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσει τις προσπάθειάς της. Συμπληρωματικό ερώτημα. Κατανοώ το ότι δεν θέλετε να συμμετάσχετε στα εθνικά πολιτικά θέματα της Βρετανίας. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με όλα αυτά τα χρέη που είναι εκτός των ισολογισμών. Εμείς έχουμε πρόβλημα με αυτό στη χώρα μας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να είναι διαφανής για όλα τα χρέη του, όπως αναμένουμε το ίδιο να κάνουν και οι τράπεζες. Αυτό σας ανησυχεί και εσάς. Απάντηση. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα όπως και άλλα θέματα που σχετίζονται με την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και στα πλαίσια των προγραμμάτων σύγκλησης και σταθερότητας. Αυτό είναι το κατάλληλο βήμα για να συζητηθούν όλα αυτά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω με τόσες λεπτομέρειες την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να μπορέσω να σας εκφράσω κατασταλαγμένη άποψη. Um, we Σας ευχαριστώ. Τέταρτος και τελευταίος γύρος ερωτήσεων. Το Λαϊκό Κόμμα πάλι κύριος Κράτσας. Κυρία Κράτσα, συγγνώμη. Κύριε Πίτροπε, τα μηνύματα για την υποστήριξη, τα μηνύματα για την υποστήριξη κρατών που βρίσκονται σε κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση όπως η Ελλάδα είναι συγκεχημένα και αντιφατικά. Η κυρία Μέρκελ υπογράμμισε την κοινή ευθύνη όλων των χωρών της Ευρωζώνης για όσα συμβαίνουν σε ένα μέλος της. Ο κύριος Ράινφελντ είπε ότι είναι εσωτερική υπόθεση της Ελλάδος και δεν αφορά κανέναν άλλον. Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Θαπατέρο είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε η Ένωση να δείξει την αλληλεγγύη της στην Ευρώπη. Ο υπουργό του κυρίου Θαπατέρο, ο κύριος Γκαρίντο, είπε ότι όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέκλεισαν κάθε περίπτωση οικονομική διάσωση της Ελλάδος. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς πώς την αντιλαμβάνεστε την αλληλεγγύη σε αυτό το τομέα. Πιστεύετε ότι είναι το ζήτημα συνδρομή σε μια χώρα με τέτοια κρίσιμη κατάσταση, πιστεύετε ότι είναι νομικό ή πολιτικό. Ευχαριστώ. You are talking to somebody who has... Uh, Κοιτάξτε, ε, μιλάτε σε κάποιον ο οποίος ε, σπούδασε ε, διεθνή πολιτική οικονομία Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ πιστεύω ότι η πολιτική και η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι η αλληλεγγύη είναι προς δύο κατευθύνσεις και προς δύο, τις δύο. Δηλαδή έχουμε μηχανισμούς όπως είναι το ε, Ταμείο Συνοχής που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να ενισχύσει κανείς την κοινωνική συνοχή και τη σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα έχουμε και κανόνες που αφορούν στη σταθερότητα, ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, όπου κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καλείται να το σεβαστεί το σύμφωνο αυτό στο πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. δηλαδή είναι αμφίδρομη η σχέση. Ε, σας είπα, εγώ θέλω να συνεργαστώ με την ελληνική κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά τελικά η ευθύνη παραμένει στην ελληνική κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο για να διασφαλίσουν ότι αυτό το υπορβολικό έλλειμμα θα κατέβει σε ανεκτό επίπεδο και επίσης τα συστημικά ε, προβλήματα στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία θα διορθωθούν. Είμαστε εταίροι, συνεργάτες, αλλά παράλληλα την ίδια στιγμή εμείς περιμένουμε οι κανόνες να γίνονται σεβαστοί. Πράγματι πρόκειται για μια πολύ σημαντική οικονομική και πολιτική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει τόσο το Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, απαντώντας στον κύριο Λάγκεν, είπατε ότι ε, στις περιπτώσεις δύσκολων συνθήκων η εκάστοτε ιδιαιτερότητα των κρατών μελών μπορεί να ληφθεί υπόψη. Ήθελα να σας ρωτήσω, στην προσπάθεια αυτή που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και που συμφωνώ απόλυτα, θα ληφθεί υπόψη το βαρύ φορτίο που έχουν για το ΑΕΠ τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι προμήθειες. Αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της ε, Ελλάδας από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. I would uh, not, not like to go into επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σήμερα το βράδυ όσον αφορά τα οικονομικά της Ελλάδας. Εκτός αυτού, ο κύριος Αλμούνια είναι ο αρμόδιος επίτροπος ε, για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα. Γιατί μιλάμε για ένα τρέχον θέμα. Τώρα, βέβαια, πιστεύω, είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα σύντομα πρόκειται να καταθέσει ένα περιεκτικό ε, πακέτο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα για να κατεβάσει το υπερβολικό έλλειμμα σε ανεκτό επίπεδο. Στην απάντησή μας τον κύριο Σλάγκεν αναφέρθηκα στους φορολογικούς ελιγμούς, το περιθώριο που υπάρχει. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτο, πολύ περιορισμένο αυτό το περιθώριο. Άρα δηλαδή η φορολογική εξυγίανση πρέπει να ξεκινήσει ταχύτατα και όχι εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε λογικό το σενάριο το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα με μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες ένα μεγάλο έλλειμμα αυτή η περίπτωση να μπορεί να ανακύψει και σε άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις κρατών μελών που σας ανησυχούν ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και από την άλλη πλευρά πώς βλέπετε τα άλλα κράτη-μέλη που είναι πιο μικρά και είναι πιο αδύναμα και μήπως πώς θα σεβαστούν τα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλει η Κομισιόν για την μείωση του υπερβολικού ελλείμματος. Απάντηση. Λυπάμαι που εστιάσαμε τόσο πολύ την προσοχή μας στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχει μη βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Όμως είναι επίκαιρη η περίπτωση. Αν κοιτάξετε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερθήκατε και σε άλλες χώρες μικρότερες και μεγαλύτεροι, ο μέσος όρος του ελλείμματος του δημόσιου τομέα αυξήθηκε από το 2008 προς το 2009 από κάτω από το 3% σχεδόν στο 7% και ταυτόχρονα Κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης, το επίπεδο του ελλείμματος αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, από το 65% στο 85%. Και στην ουσία χάνουμε τα όσα είχαμε επιτύχει τα τελευταίες δύο δεκαετίες εξαιτίας αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό σας δείχνει και την κλίμακα των προκλήσεων και δείχνει το πόσο ζωτική σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό τώρα, έγκαιρα και όχι να το αφήσουμε για όταν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μια αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και μια ενίσχυση της εποπτείας των κρατών και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτόν τον μεγάλο στόχο. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι η περίπτωση της Ελλάδος δεν είναι μοναδική. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ, σας ανησυχούν άλλες περιπτώσεις κρατών μελών και θα ήθελα να κατανοήσω τι μέτρα προτείνεται, συστήνεται στα άλλα κράτη ώστε η περίπτωση της Ελλάδος να μην επαναληφθεί σε άλλα κράτη-μέλη. Yes, Απάντηση. Ανησυχώ για τις τάσεις των δημοσίων οικονομικών σε πολλά άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα, στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς στιγμήν έχουμε τάσεις μη βιώσιμες για το έλλειμμα και το χρέος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τώρα να αναλάβουμε δράση. Και η καλύτερη συνταγή για όλα τα κράτη-μέλη και για την Ευρωζώνη είναι να σεβαστούν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έγκαιρα να λάβουν αποφάσεις για την φορολογική εκαθάριση, να αναμένουν να εξυγιανθεί η οικονομία τους και πολύ προσεκτικά να αξιολογήσουν κάθε γραμμή του προϋπολογισμού τους για να βελτιώσουν την ποιότητα των δημοσίων τους οικονομικών για να έχουμε μεγαλύτερη αξία για τα χρήματα που ξοδεύουμε. Ε, Μίτσελ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Φανρομπάη στη Γερμανία πρόσφατα είπε ότι πρέπει να σταθμίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη 2% αν θέλουμε να βγούμε από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά. Πέρα από την ανάλυση δηλαδή στο Κοινοβούλιο που λέμε ότι έχουμε δυσκολίες, πώς θα αποφύγουμε να επανέλθουν τέτοιες δυσκολίες. Δεν πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και εσείς τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Τι εννοείτε recalibration στα αγγλικά. Αυτό που σας ζητάω είναι τι εννοεί ο κύριος Φανεροπάη όταν χρησιμοποιείς αυτόν τον όρο recalibration. Δεν το ξέρετε. Ε, τι εννοούσε. Και τι θα κάνει η Επιτροπή για να στηρίξει τις προτάσεις αυτές. Αυτό που λέει ο κύριος Φανρομπάου είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ανάπτυξη 2%. Αλλιώς είναι πολύ σκοτεινό το μακροπρόθεσμο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο από κοινού να μπουν σε μια διαδικασία ώστε να πετύχουν αυτό που ο κύριος Φανροπάη ονομάζει recalibration. Ε, κοιτάξτε, εντάξει, είναι και θέμα γλώσσας που χρησιμοποιεί κανείς. Σίγουρα θα κοιτάξουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και είτε μιλάμε για recalibration είτε μιλάμε για αναζωγόνηση της οικονομικής ανάπτυξης, το ίδιο είναι. Ο κύριος Φανρομπάου μιλάει εκ μέρους του αυτού του και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως πρόεδρος. Εγώ μιλάω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα οικονομικά και νομισματικά ζητήματα, εφόσον βέβαια επιβεβαιώσετε τη θέση μου σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και αναλάβω τα καθήκοντά μου. Είναι πολύ ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη η συζήτηση σήμερα το βράδυ επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη, στην απασχόληση επίσης και στο γεγονός ότι πρέπει να καταφέρουμε καλύτερα να πετύχουμε υψηλό δυναμικό υπέρ υγιών ε, δημοσίων οικονομικών, ώστε να στηρίξουμε τη στρατηγική μας για την Ευρώπη του 2020 με μια δυνατή οικονομία, καινοτομία, εκπαίδευση και άλλους παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί για την οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και εννοείται ότι δεν ευθύνεται αυτός για τόσα λέει ο κύριος Φανερομπάου. Αλλά θέλω να το ρωτήσω. Συμφωνείτε ότι με νέο κοινοβούλιο, νέο συμβούλιο, νέα επιτροπή έχουμε τώρα μια νέα ευκαιρία για να προχωρήσουμε με την ανάκαμψη και να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αντί να κοιτάμε πίσω να κοιτάμε προς τα μπρος. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν πήγαν όλοι άσχημα με αυτή την οικονομική κρίση. Ορισμένοι τα κατάφεραν με τις αποταμιεύσεις τους. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή σαν σημείο νέας εκκίνησης. Απάντηση. Ναι, σίγουρα και πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάκτηση εμπιστοσύνης. Σε κάθε επίπεδο. Γιατί αυτή βοηθάει να υπάρξει νέος δυναμισμός στην Ευρώπη. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι η ανάπτυξη, δηλαδή πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε να υπάρξουν επενδύσεις υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και να ενθαρρύνουμε και το τραπεζικό τομέα ώστε να υπάρχουν πιστώσεις και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις και συγχρόνως στο δημόσιο τομέα πρέπει επίσης να δουλέψουμε προκειμένου να έχουμε υγιή δημόσια οικονομικά. Είναι λοιπόν διτή η πρόκληση. Αυτή την πρόκληση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σίγουρα χρειάζεται αποφασιστικότητα από την πλευρά μας και στις δύο πτυχές του διδήμου αυτού. Ανάπτυξη δηλαδή και υγιή δημόσια οικονομικά. Ευχαριστώ. Σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Φέλλερ τώρα. predsednica. Πρόεδρε. Κύριε Ρέιν, κατά τη διάρκεια των διακοπών ανασάναμε. Ε, δεν συζητήσαμε για ε, την ύφεση, ε, συζητήσαμε περισσότερο για το χιόνι, αλλά η κατάσταση παρέμεινε ίδια. Στην Ευρώπη ε, πάρα πολλές ε, εταιρείε έκλεισαν, χάθηκαν θέσεις εργασίας, ε, καταστράφηκαν όνειρα. Από κοινωνική και οικονομική άποψη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι καθοριστική σημασίας. Μιλάμε για 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 99% αυτών είναι ε, μικρομεσαίες. Είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα γραφειοκρατίας, προβλήματα στην πρόσβαση σε κονδύλια. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, πώς προτίθεστε να διευκολύνετε την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάλα για αυτή την ε, ερώτηση που με αγγίζει πάρα πολύ γιατί και εμένα ο πατέρας μου ήταν ε, επιχειρηματίας και μιλάτε σε ε, γιο επιχειρηματία, αυτοδημιούργητο, ο οποίος έχει συστήσει μία μικρή επιχείρηση ανταλλακτικών. Εκεί πέρασα τα χρόνια μου όταν ήμουν νέο, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί ενδέχεται να δει ότι παραβίασα και εγώ του κανόνε περί παιδική εργασία. Αυτά. Όσον αφορά τώρα την ε, οικονομική ανάπτυξη, πράγματι πρέπει να δούμε λιγάκι όλα τα θέματα που επηρεάζουν τις, ε, ε, τη μελλοντική λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να βρούμε πρόσβαση, τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων αυτών επιχειρήσεων σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Και ως εκ τούτου, πολλοί έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον τραπεζικό τομέα. Ε, τώρα δεν είναι η εποχή των ε, μεγάλων ε, πριμ και των μεγάλων μερισμάτων. Το πρόβλημα είναι να είναι ισοσκελισμένοι οι προπολογισμοί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις πράγματι πρέπει να διευκολυνθούν έτσι ώστε αυτή η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας να μπορέσει να ανακάμψει και να ε, καλύψει τις προσδοκίες μας όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το σκέλος της απάντησης. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι χρηματοψηφιακές αγορές καταστράφηκαν από την οικονομική κρίση και τα ε, κυριότερα θύματα ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα ε, πρόσβαση σε κονδύλια. Ε, χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα των αφορολογουμένων για να διασωθούν οι τράπεζες, οι οποίες τώρα από την πλευρά τους δεν ε, δανειδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας, ε, κατόπιν του, του ε, αύξηση της ανεργίας, λιγότερες επενδύσεις, ε, μικρότερη εμπιστοσύνη. Μήπως έχετε κατά νου συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε πραγματικά να διευκολύνετε τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Ταγιάννη, τον Αντιπρόεδρο ο οποίος ε, είναι αρμόδιος ε, για τη βιομηχανία και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Ταγιάννη λοιπόν θα ασχοληθεί κυρίως με θέματα που έχουν σχέση με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και παράλληλα, όταν θα εξετάσουμε τα κοινοτικά εργαλεία που υπάρχουν για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, θα λάβουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ότι τα περισσότερα κονδύλια προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή από τις τράπεζες και άλλα ε, πιστοτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ροή κεφαλαίων θα φτάνει στο στόχο της, θα φτάνει στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και παράλληλα Οφείλουμε να αξιολογήσουμε τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα το επιχειρηματικό καινοτόμο κεφάλαιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Ρέν, ο Βρετανικός τύπος και κάποιοι βουλευτές φοβούνται ότι η σταθερότητα του ευρώ έχει υπονομηθεί εξαιτία περιπτώσεων όπως αυτή της Ελλάδος με τα μεγάλα ελλείμματα. Σημερίζεστε αυτή την ανησυχία και αν ναι, προβλέπετε να εφαρμοστούν οι οικονομικές κυρώσεις που προβλέπονται στο σύμφωνο σταθερότητας ή μήπως πιστεύετε ότι η σταθερότητα του ευρώ οφείλεται στο οικονομικό βάρος όλη της όλης της Ευρωζώνης που είναι πολύ μεγαλύτερη από τα συστατικά στοιχεία της Ευρωζώνης. Μήπως υπερεκτιμούμε την επίπτωση της ελληνικής κατάστασης πάνω στο ευρώ. Ε, πριν από μερικά χρόνια η πόλη της Νέας, Ευρω... Ε, Υόρκης ήταν σε χρεοκοπία και αυτό δεν επηρέασε το δολάριο ακόμα και αν το ΑΕΠ της Νέας Υόρκης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδος. Απάντηση. Ναι. Θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να σεβαστούν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τις ρήτρε του για το υπερβολικό έλλειμμα. Είναι σημαντικό για τις ίδιες τις χώρες, τους πολίτες τους και σε συστημικούς, για συστημικούς λόγους για την ζώνη ευρώ. Και γι' αυτό εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, γιατί αυτό υπονοεί ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μακροοικονομική του σταθερότητα και τα δημόσια του οικονομικά είναι υγιή και βιώσιμα. Αυτό προς όφελος της ίδιας της χώρας αλλά και προς όφελος συνολικά της Ευρωζώνης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε πολλές χώρες και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει το εάν οι επόμενες αποφάσεις στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβαλλικού ελλείμματος θα ληφθούν από την Κομισιόν τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Με άλλα λόγια, το εάν ο Επίτροπος που θα παρουσιάσει την απόφαση θα είναι ο Χωακή Μαλμούνια ή εγώ ίδιος εάν επιβεβαιώσετε την θέση μου συμπληρωματικό ερώτημα. Κύριε Επίτροπε, φοβάστε για τη σταθερότητα του ευρώ εξαιτία τη Ελλάδος ή και δεύτερο ερώτημα, θα εφαρμόσετε τι οικονομικές κυρώσει που προβλέπει το σύμφωνο ή συμφωνείτε και εσείς ότι αυτό, όπως είπε και ο κύριος Λαμπή, είναι ο μεσαιωνικός χαρακτήρας από του Συμφώνου Σταθερότητα, ότι δεν μπορεί δηλαδή να υποβάλουμε οικονομικέ χειρώσει σε κάποιον που είναι ήδη αδύναμο. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα με την Ελλάδα και το υπερβολικό έλλειμμα και χρέος είναι πολύ σοβαρό. Ιδιαίτερα για την ίδια την Ελλάδα, για τους Έλληνες πολίτες φορολογούμενους, αλλά επίσης έχει και δυνατότητα επιρροής σε όλη την Ευρωζώνη. Δεν είναι τόσο σοβαρό ακόμα που να απειλήσει την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Γι' αυτό είναι απόλυτα επίγον η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική βουλή να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα με απτά μέτρα για το σύμφωνο σταθερότητας και τις, ε, τα εργαλεία που διαθέτει. Εάν με επιβεβαιώσετε ως Επίτροπο, δεν αποκλείω οποιαδήποτε χρήση εργαλείου που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά τώρα πρέπει να ληφθεί γρήγορη δράση για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης. και να έχουμε εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε υγιή δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ρεν μπορεί να μιλήσει την πέμπτη του γλώσσα τώρα. Σουηδικά. Λοιπόν, όταν η Σουηδία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995, δεν διαπραγματευτήκαμε τίποτα εξαιρέσει για το πώς θα προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία όμως έχουν εξαιρέσει. Ρωτάω λοιπόν τον ελπίζω μελλοντικό επίτροπο και είναι ένα λεπτό ζήτημα για μας στη Σουηδία. Το ερώτημά μου έχει ως Μπορεί η Σουηδία στο μέλλον να συνεχίσει να βρίσκεται εκτός Ευρωζώνης χωρίς να κινδυνεύει να μην αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα. Εσείς αυτό το θέμα θα το συζητήσετε με τη Σουηδική Κυβέρνηση. Θα συζητήσετε τις απόψεις που υπάρχουν για ε, να ενταχθεί όχι στην Ευρωζώνη η Σουηδία. Απάντηση. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που είναι σημαντική για τη Σουηδία αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η Σουηδία δεν διαπραγματεύτηκε για εξαιρέσει όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην όταν ήρθε στους κόλπους μας. Και εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν η Σουηδία έκανε το δημοψήφισμά της το 2003 για να ενταχθεί στην Ευρωζώνη όχι και ξέρουμε όλοι ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος. Όλο αυτό μας έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση, μια πραγματικότητα και είναι γεγονός ότι το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί στον σουηδικό λαό καταρχήν. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης, είμαι από μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης και πολύ θα ήθελα η Σουηδία να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο ίδιος ο Σουηδικός λαός. Πρόσφατα Είδα ε, μια συνέντευξη με τον ε, Σουηδό Υπουργό Οικονομικών, τον Άντερ Πολ, που δημοσιεύθηκε σε μια σουηδική εφημερίδα. Στη συνέντευξη αυτή λοιπόν ο Άντερ Πολ μίλησε για την σημασία που έχει για τη Σουηδία να μπορεί να παίρνει πλήρως αποφάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από την Ευρωζώνη. Και αυτό είναι ένα καλό σημείο κίνησης για τη συζήτηση. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι ευχαρίστως να, να συμμετάσχω σε συζητήσεις για αυτό το θέμα, αλλά σέβομαι απόλυτα τα δικαιώματα του Σουηδικού λαού να αποφασίσουν για αυτό το θέμα. Συμπληρωματική ερώτηση. Σε δημοσκοπήσεις που έγιναν πρόσφατα στη Σουηδία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στην Ευρωζώνη της Σουηδίας. Ορισμένοι λένε ότι η αστάθεια διακυμάνσεις που είχαμε και που έχουμε στις νομισματικές συναλλαγές είναι πράγματα τα οποία ανησυχούν τον κόσμο στη Σουηδία. Πολλοί λοιπόν είπαν ότι όταν ε, έπεσε πριν από λίγα χρόνια κατά 25% η κορώνα, αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Οπότε κύριε Ρεν, εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό, να εξετάσετε το θέμα αλληλεγγύης. Στο κάτω-κάτω από την Φιλανδία είσαστε εσείς. Δεν θα έπρεπε σαν έδειξη αλληλεγγύης προς τη Σουηδία να βοηθήσετε για την ένταξή μας στην Ευρωζώνη. Απάντηση. Κοιτάξτε, θα επαναλάβω λίγο αυτά που είπα και πριν. Δηλαδή ότι είναι θέματα που συζητιούνται στο εσωτερικό της Σουηδίας, είναι θέμα δηλαδή εσωτερικής πολιτικής και δεν θα ήθελα να αναμειχθώ. Δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε δηλαδή αν εγώ ξεκινούσα να υιοθετώ ε, θέσεις και να τοποθετούμε όσον αφορά τα εσωτερικά ζητήματα της Σουηδίας. Εγώ θα προτιμούσα η ίδια η Σουηδία και ο Σουηδικός λαός να συζητήσουν με οριμότητα το θέμα αυτό και μετά κάποια στιγμή ελπίζω να ληφθεί σχετικά και μία απόφαση. Είμαι και εγώ από τη Βόρεια Ευρώπη και πολύ θα ήθελα να δω τη Σουηδία να συμμετέχει στην Ευρωζώνη. Γιατί έτσι συμπληρώνεται, αν θέλετε, το παζλ της Βόρειας Ευρώπης μέσα στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Στην ώρα μας. Τελειώσαμε με τις 32 ερωτήσεις και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην τελική τοποθέτηση του προτινόμενου επιτρόπου. Προηγουμένως όμως θέλω να υπενθυμίσω τα τρία σημεία τα οποία έθεσα και στην αρχή της συνάντησης αυτής. Σας τα έχω δώσει και γραπτά. Πρόκειται για την συνεργασία που θα έχετε με την Επιτροπή μας, με τα έγγραφα τα οποία θέλουμε και την ενημέρωση που θέλουμε να έχουμε έγκαιρα από εσάς. Να μας μιλήσετε για τη συνεργασία των τριών επιτρόπων που ασχολούνται με θέματα που εξετάζει και η Επιτροπή μας και να μας μιλήσετε λίγο και για τις ε, ρυθμίσεις στο δημοσιονομικό σύστημα. Παρακαλώ λοιπόν για την ε, τελική σας τοποθέτηση, κύριε Ρεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπα και στην αρχή, ε, δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την Επιτροπή σας. Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω για γνωστά και άγνωστα θέματα. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορώ να υπογραμμίσω, γιατί το θέμα είναι αν δεν γνωρίζω τι συμβαίνει σε μία περίπτωση, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορώ να το αποκαλύψω. Αυτό θα είναι μια πραγματική πρόκληση. Ε, θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές όλες οι προκλήσεις. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό που παίρνω από αυτή την ουσιαστική συζήτηση γεμάτη από ρεθίσματα, ε, υποβάλλατε σκληρές ε, ερωτήσεις επί της Σωστά πράξατε. Κατά την άποψή μου, η ακρόαση αυτή απέδειξε το ότι έχουμε κοινούς στόχους που είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική, κοινωνική ευρωπαϊκή οικονομία. Και η συζήτηση επίσης ε, κατέδειξε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει να υπάρχουν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Πιστεύω εξάλλου ότι από την ανταλλαγή απόψεων κατέστη σαφές ότι τρεις είναι οι στόχοι που θεωρούνται οι σημαντικότεροι και επικράτησαν σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να εργαστούμε για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ανατάξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία κινητοποιώντας όλους τους παράγοντες ε, για να υπάρχει μια πράσινη οικονομική ανάπτυξη. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να ενισχύσουμε το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, να συμπεριληφθούν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πολιτική 2020 πρέπει να στεφθεί από επιτυχία και νομίζω αν πράξουμε αυτά που ανέφερα θα επιτύχουμε αυτό το στόχο. Οφείλουμε να ενισχύσουμε τα θεμέλια των οικονομιών μας ενισχύοντας τα δημόσια οικονομικά, γιατί μόνο με υγιή δημόσια οικονομικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ε, την ανεργία και το μέλλον. Και τέλος πρέπει να βελτιωθούμε στο να προάγουμε τα κοινά μας συμφέροντα, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη που είναι να ενισχύσουμε την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν είμαστε ενωμένοι προς τα έξω θα μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή, να ε, προβάλλουμε περισσότερο το, κύρο μας, το κύρος μας με συγχωρείτε, στα παγκόσμια οικονομικά. Κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση επέφερε μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Προέκυψε ανθρώπινο κόστος με την έννοια της ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε συγκεκριμένες αποφασιστικές ενέργειες για να μην διακινδυνέψουμε ένα κομμάτι αυτής της ζημιάς να μετατραπεί σε μόνιμη. Οι πολίτες Ευρώπης περιμένουν η Ευρώπη να τους προσφέρει και γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμεθα να ικανοποιήσουμε αυτές τις ε, προσδοκίες τους. Εγώ προσβλέπω σε εσά, προσβλέπω στη στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας και δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος αυτής της μεγάλης πρόκλησης που είναι η βελτίωση των οικονομικών και να επανέλθει η Ευρώπη στο δρόμο της ανάπτυξης και της ε, βιώσιμης ανεργίας. Αυτά θα τα καταφέρουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ και όπως σας είπα ελπίζω να έχουμε και στο μέλλον συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Προτινόμενο Επίτροπο και όλους τους Ευρωβουλευτές που τήρησαν τον χρόνο τους. Η συνάντηση αξιολόγησης θα λάβει η χώρα σήμερα το βράδυ, 8 με 9, στο ASP 1G3 είναι συνάντηση ανοιχτή συντονιστών που σημαίνει ότι μπορούν να έρθουν και προβουλευτές και προσωπικό, όχι βοηθή και εννοείται όχι δημοσιογράφοι ή κοινό. Στην ΑΣΠ 1G3 κλείνει η συνάντηση αυτή στις 8, στις 8.